Ich Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. So, schönen guten Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε και κύριοι. Καταρχήν, οι αποφάσει των συντονιστών από την χθεσινή συνεδρίαση. Σα έχουν διανεμηθεί τα αντίγραφα και αν δεν ε, υποβληθούν ενστάσεις μέχρι σήμερα το μεσημέρι στι 1 θα θεωρούνται εγκεκριμένε και, αυτά, και αυτά του, της 25ης Ιανουαρίου. Και τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία για την ε, απαλλαγή της Επιτροπής και των οργανισμών. Καταρχήν θα ελέγξουμε το σύστημα. Άρχεται η ψηφοφορία.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 have Ο εισηγητή είναι ο κ. Μασιμιλιάνο Σαλίνη και προχωράμε στην τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πίτερ Λούντκριν. 13 υπέρ. Voting list, Σχέδιο γνωμοδότησης για την, για την απαλλαγή του Γενικού Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. David, 13 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 46 υπέρ 37 ε, κατά μία εποχή εγκρίνεται. Τώρα θα περάσουμε στη ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροπορίας. Η Νέσα Γιάλα Σάντερ είναι η συγγήτρια. Τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ, συγγνώμη, έξι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και εδώ υπάρχει μια προφορική τροπολογία στην τροπολογία 5 της κυρία Σάντερ. Thank It's uh, in the fields Στους τομείς της ασφάλειας για, την, ε, ε, για τις κοινωνικές, έχουμε συμπεριλάβει στην τροπολογία τις ε, κοινωνικές προϋποθέσεις και το περιβάλλον. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία της κυρίας Έντερ. Ωραία, δεν την ψηφίζουμε λοιπόν. Πάμε στην 5 χωρί την προφορική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Τροπολογία 7. Υπέρ. Όχι, 4. 4, 4. Τροπολογία 4. 4 Κατα Καταπίπτει 4. Άρα την 7. Τροπολογία 7 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. 41 ψήφοι υπέρ, 4 κατά και 1 αποχή. Εγκρίνεται. Επόμενη ψηφοφορία. Πάμε στο ΣΕΖΑΡ. Κοινή επιχείρηση ασφάλεια τη αεροναυτιλίας. Η κυρία Ενέσα Γιώλα Σέντερ είναι η συγγήτρια. Και πάλι. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία.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 14 υπέρ, 29 κατά, 3 αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 12 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 39 ψηφί υπέρ, 6 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Πάμε στην τελευταία ψηφοφορία για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Και πάλι η συγγετρία η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Κατά. Τι. Έχουμε μια προφορική τροπολογία. Κυρία Σέντερ. Την παράγραφο 3 συμπεριλαμβάνουμε σύμφωνα με τις δημοσιονομικές ε, αρχές στα πλαίσια του MFF. Ότι πρέπει δηλαδή ο προπολογισμό να ε, εμπίπτει μέσα στο ε, MFF. Υπάρχουν αντιρρήσει. Όχι. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 1 με την προφορική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Η ένα καταπίπτει γιατί έχει οθετηθεί η προφορική τροπολογία. Πάμε στη 2. Αυτό είπα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 17 υπέρ, 29 ψήφι κατά, καμία αποχή. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, απορρίφθηκε είπαμε, 9 υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε στην προφορική τροπολογία και πάλι της κυρίας Σέντερ, παρακαλώ. Πάλι στα αγγλικά. Προσθέτουμε στο τέλος και έχει ε, δημιουργήσει ε, επιπλέον ελέγχους για να παραμείνουν ε, εφόσον υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι γίνονται οι έλεγχοι με αποτελεσματικό τρόπο. Είναι έτσι ένας τρόπος να δώσουμε μια απόχρωση στο, στο κείμενο του εισηγητού. Ε, υπάρχει αντίδραση για αυτή την προφορική τροπολογία? Όχι. Ωραία. Οπότε ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία 2. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά πάμε στη 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Abstimmung ist geschlossen. Πέρα ψηφοφορία. 37 ψήφοι υπέρ, 9 ψήφοι ε, κατά, καμία αποχή εγκρίνεται και θερμά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Τελείωσαν λοιπόν οι ψηφοφορίε μας. I ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Wir kommen nun zu dem nächsten Punkt. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μακάου σχετικά με ορισμένες σχετικά με ορισμένες των αεροπορικών μεταφορών. Η συγητή συνοντείται Λέμπρεχτ Κόχ και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ να σας παρουσιάσω την, ε, το ακριβές μου σχέδιο για μια συμφωνία μεταξύ της, του Μακάου, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και και θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, πρόκειται για μια συμφωνία με την οποία οι 15 διμερείς ε, συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μακάο θα αντικατασταθούν. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία δεν είναι επίμαχη και στην οποία έγιναν κάποιες βελτιώσεις και αλλαγές ούτως ώστε να υπάρξει συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ιδιαίτερα όσον αφορά το δίκαιο ανταγωνισμού, πτυχές ασφαλείας, φορολογικά ζητήματα και την ελευθερία εγκατάστασης και με όλα αυτά εκπληρώνουμε τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η συμφωνία ήδη ε, ε υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2013, ωστόσο ε, χρειάζεται η συμφωνία του, η έγκριση του Κοινοβουλίου για να τεθεί σε ισχύ. Εμείς ως Κοινοβούλιο δεν θα υποβάλουμε τροποποίηση, δεν ε, μπορούμε να υποβάλουμε μόνο τροπολογίες οι οποίες αναφε, στηρίζονται στη δική μου σύσταση και εγώ επειδή η έκθεση δεν παρουσιάζει προβλήματα σας ε, συστήνω να την υπερψηφίσετε. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ε, εδώ παρεμβάσεις. Γκεζίνε παρακαλώ. Θα μπορώ να πω ότι στηρίζω την έκθεση ε, εξ ονόματος του σκιώδου συζητητού Χωσέ Ιγνάσιο Μαρία. Ευχαριστώ. Φώστερ. E ναι, εκ μέρου του ΕΣΥΑΡ e ευχαριστούμε τον εισηγητή για την δουλειά του και στηρίζουμε την θέση του. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Δεν ξέρω η Κομισιόν μήπως θέλει το λόγο. Όχι. Ωραία. Άρα, η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες, για να είναι έτσι πιο τυπικά τα πράγματα, 24 Φεβρουαρίου μέχρι τις 12 ε, το μεσημέρι και η, μόνη τροπολογία είναι να αρνηθούμε ουσιαστικά, να απορρίψουμε την ε, συμφωνία. Δεν μπορούμε να υποβάλουμε, δεν επιτρέπονται άλλες, άλλου είδους τροπολογίες. Κλείνουμε λοιπόν το σημείο αυτό της σημερινής διάταξης και πάμε στο επόμενο. Έλεγχος. Προετοιμασία πράξης κατεξουδότηση για την ε, παροχή σε επίπεδο ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις. Να δώσουμε τον ε, λόγο στην ε, Κομισιόν, στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, για 10 λεπτά το πολύ. Δεν είναι κανείς εδώ? Α, πολύ ωραία. Mm-hmm. Yeah. Gut, dann Να δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια τότε. Η Γκεζίνε Μάισνερ είναι η εισηγήτρια. Ναι, αλλά εγώ θέλω να έχουμε και την Κομισιόν εδώ. Αλήθεια, σοβαρά σας το λέω. Γιατί σε αυτή τη διαδικασία είναι απαραίτητο να είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω να το αλλάξουμε, αλλά μετά έχουμε το ακρόαση το απόγευμα. Για το επόμενο σημείο που πάλι έχουμε ανακοίνωση της Επιτροπ... ε, παρουσίαση από την Επιτροπή, είναι εκπρόσωπος Κομισιόν εδώ. Για την, ανταλλαγή ηλεκτρονικών, ε, για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών. Ούτε για αυτό το θέμα είναι κάποιος εδώ. I must say that it's the first time. Πρωτοφανές που συμβαίνει κάτι τέτοιο στα 12 χρόνια. Okay, then I think we make a rest until 10 o'clock. Κάνουμε ένα διαλυματάκι λοιπόν μέχρι τις 10 και βλέπουμε μετά.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 I think now we will start. Θα ξεκινήσουμε τώρα. Εδώ είναι η Κομισιόν, αλλά λείπουν πολλοί από εμά. Hello, Roberto. No, Michele. Michele. Roberto και Michele καθίστε. Okay, then we continue and the floor is yours. Συνεχίζουμε η κυρία Επίτροπος. Δεν είμαι Επίτροπος. Είμαι από την DigiMove. Θα ήθελα καταρχάς βέβαια να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι εδώ σήμερα. Γιατί, γιατί αυτό το θέμα μας μας απασχολεί εδώ και καιρό Σε όλες τις συζητήσεις είχαμε την συμμετοχή της γραμματείας της ΤΡΑΝ. Οπότε χαίρομαι που είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω το που βρισκόμαστε σε σχέση με την εκπόνηση κατά της νομοθεσίας για αυτό το θέμα. Ομονοούμε νομίζω σε αυτό το θέμα. Μεζόμαστε τους ίδιους στόχους και πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα να θυμόμαστε ότι το θέμα αυτό δεν είναι νέο για την Κομισιόν. Ήδη προβλεπόταν στη Λευκή Βίβλο το 11 για τις μεταφορές. Πέρασε πολύς χρόνος από τότε και θα σας εξηγήσω σε λίγο το τι κάνουμε. Πιο πρόσφατα εθετήσαμε ένα γράφο εργασία της Κομισιόν με ένα λεπτομερή οδικό χάρτη για τον σχεδιασμό των μεταφορών και τα εισιτήρια. Επίσης είχαμε και μια γνωμοδότηση πρωτοβουλίας από το Κοινοβούλιο σε σχέση με τις ολοκληρωμένες μεταφορές. Υπάρχουν λοιπόν υπάρχει μεγάλη πολιτική υποστήριξη σε αυτόν τον τομέα. Θα μιλήσω για αυτή την κατουσιοδότηση νομοθεσία η οποία σχετίζεται άμεσα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker. Μιλάμε για τη στρατηγική της ε, ψηφιακής κοινωνίας, την Ενεργειακή Ένωση. Πράγματα δηλαδή που θα μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε αυτή τη βιώσιμη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Ανάπτυξη, απασχόληση, ε, ένα στο μέσο που έχουμε μεγάλο δυναμισμό των επιχειρήσεων και ενή αγορά. Η διδραστικότητα είναι από τα κύρια κριτήρια λοιπόν ώστε αυτές οι υπηρεσίες να λαμβάνουν χώρα πανευρωπαϊκά. Αλλά ταυτόχρονα να ωφελούνται και να κερδίζουν επιχειρήσεις από αυτό το πλαίσιο. Τι έχει γίνει λοιπόν. Ό,τι έχει γίνει, κυρίως έχουν γίνει λόγω Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Στο τέλος του 8, να θυμηθούμε ότι υπέβαλε μια πρόταση η Κομισιόν και ζήτησε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο από την Κομισιόν να διευρύνουν αυτή την οδηγία και να δουν τη διάδραση με άλλους τρόπους μεταφορών. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα του δικού σας αιτήματο, που ήταν πολύ σωστό τότε να μας παροτρύνετε να σκεφτούμε περισσότερο και εναλλακτικά. Κάποια στοιχεία. Μια εξωτερική μελέτη μας βοήθησε να εξετάσουμε εδώ τους όγκους για τους οποίους συζητάμε εδώ. Έχουμε 3 εκατομμύρια διασυνοριακές μετακινήσεις στην Ένωση. Δεν μόνο για αυτούς που το κάνουν καθημερινά για την εργασία τους. Αυτό δείχνει τη σημασία που έχει αυτό το θέμα για τους πολίτες. Έλεγα ότι συμμεριζόμαστε τους ίδιους στόχους όλοι αυτό που θέλουμε είναι το να υπάρχει πλήρης κάλυψη και πλήρης ενημέρωση για τους πολίτες με εκτενείς πληροφορίες για τα ωράρια των μετακινήσεων που θα καλύπτει όλους τους τρόπους, όλα τα μέσα ταξιδιού και μεταφορών. Θα πείτε κάποιοι από εσά, εντάξει, αν σχεδιάσω το ταξίδι μου σήμερα, ήδη μπορώ να κάνω πολλά. Δίκιο έχετε, αλλά παρόλα αυτά και τώρα νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή για να χρησιμοποιήσουμε τις διαφάνειες εδώ στην οθόνη τη μεγάλη. Όταν θέλουμε να κάνουμε μια διασυνορική μετακίνηση από το α στο β, κοιτάμε πούμε την απόσταση μεταξύ δύο πόλεων. Είναι πολύ πιο δύσκολο αν προσπαθήσουμε να διαργωνώσουμε το ταξίδι μας, όχι μόνο σε σχέση με την άφηξη σε ένα αεροδρομικό σταθμό ή σε ένα αεροσταθμό, αλλά μέχρι και το τελευταίο μίλι Υπάρχουν λοιπόν διάφορα μοντέλα, όπως βλέπετε εδώ στην οθόνη. Το πρώτο είναι αυτό της αποκεντρωμένη προσέγγισης. Έχουμε αυτό το σχεδιασμό ταξιδιού με διάφορα μέσα μεταφοράς που παρέχεται από ένα μεγάλο πάροχο. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω αντανακλά την παροχή από ιδιώτες όσον αφορά το ταξίδι. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να καλύψουμε την αναχώρηση και την τελική άφηξη, τότε θα πρέπει να βασιστούμε σε πολύ λεπτομερέστερο επίπεδο πληροφοριών. Αυτά δηλαδή που παρέχονται στο εσωτερικό μιας πόλης. Εδώ βλέπετε λοιπόν το απακεντρωμένο μοντέλο. Το αριστερό σας δείχνει ότι υπάρχει η μεγάλη απόσταση, διασύνδεση και υπηρεσίες. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και αυτό το κίτρινο σημείο όπου εκεί πραγματικά βασιζόμαστε σε πληροφορίε οι οποίε παρέχονται σε τοπικό αστικό επίπεδο. Θα ρωτήσετε τώρα. Γιατί λοιπόν αυτή η ανάλυση ήταν χρήσιμη στην εκπόνηση της δουλειά μας. Ήταν πολύ χρήσιμη να σου την αλήθεια στο να κατανοήσουμε τι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην κατεξοδότηση νομοθεσία, ώστε να στηρίξουμε έναν πανευρωπαϊκό σχεδιασμό ταξιδίου. Να σας πω ότι εμείς και οι πελάτες δεν διαφορμάστε τόσο πολύ για τις πληροφορίες που παρέχονται, ας πούμε, στην πρώτη λύση ή τη δεύτερη ή την τρίτη επιλογή. Αυτό τελικά δεν έχει τόσο σημασία. Όταν συζητήσαμε λοιπόν με τους εμπειρογνώμονες από τις χώρες μέλη. Και ήδη πολλά συμβαίνουν στις διάφορες χώρες μέλη πάνω σε αυτό το θέμα και εξελίσσεται γρήγορα, όπως είδαμε στις συζητήσεις με τι χώρες μέλη. Προσπαθήσαμε λοιπόν να καταλάβουμε το εξής. Αν εξετάσουμε χώρες σαν την Αυστρία ή την Τσεχία, που ήδη έχουν ένα εθνικό σχεδιασμό ταξιδίου με διάφορα μέσα. Αν έχουμε λοιπόν ένα νέο μοντέλο το οποίο βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στους χρήστες για την κινητικότητα ας πούμε. Αν δούμε τη Γαλλία. Είχαμε πρόσφατα ένα νομοσχέδιο που πραγματικά προβλέπει την διάθεση δεδομένων Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται προσπάθειες να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν όσον αφορά τη διάθεση αυτών των ε, στοιχείων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα στοιχεία και προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε διάφορους τρόπους πολυτροπικού ταξιδιού. Κοιτάξαμε ας πούμε τη φύση του ταξιδιού, κοιτάξαμε ας πούμε τα ωράρια. Αλλά το κάναμε αυτό με βάση μια λειτουργικότητα η οποία εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Είδαμε α πούμε τι υπηρεσίε. Βλέπουμε εκεί στα διάφορα σημεία ότι πράγματι μπορούμε να συνδέσουμε τι διάφορε υπηρεσίε που παρέχονται. Οπότε την ίδια προσέγγιση που είχαμε σε προηγούμενες κατεξοδότηση νομοθεσίες, κάναμε το ίδιο. Δηλαδή ζητήσαμε από τι χώρε μέλη να δημιουργήσουν κάποια σημεία, να έχουν μια προσέγγιση βαθμιαία, όπου θα διευρύνουμε το γεωγραφικό πεδίο με στόχο βέβαια να καλύψουμε τα πάντα στο δίκτυο. Τη βασική μετακίνηση και όλες τις υπόλοιπες επεκτάσεις της. Είχαμε την έκθεση του κυρίου Κόχ βέβαια. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε όλο το δίκτυο μέχρι το 2023. Θα απαντήσω στην συνέχεια σε ερωτήσεις σας, αλλά να σας πω ότι και πάλι μιλάμε για μια κατεξουσιοδότηση πράξη, η οποία δεν καθιστά υποχρεωτική την πρόσβαση στα δεδομένα, αλλά όταν τα ψηφιακά δεδομένα αυτά θα είναι διαθέσιμα, τότε θα πρέπει σε τυποποιημένη μορφή να είναι διαθέσιμα αυτά σε εθνικό επίπεδο. Είχαμε τεράστια ανάπτυξη Εντάξει, στην αεροπορία το ξέρουμε. Στο σιδηρόδρομο επίση και στο τομέα των δημοσίων μεταφορών. Τα πράγματα προχωράνε τόσο γρήγορα που πολύ σύντομα νομίζω θα είμαστε σε θέση να παράσχουμε συνολικές δεξιωτικέ πληροφορίε στους πολίτες και να θέσουμε την βάση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα εισιτηρίων σε κάποια στιγμή στο μέλλον. Νομίζω ότι είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και μέσω των απαντήσεων θα, θα συμβάλλω περισσότερο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μάισμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και για την ε, έκθεση. Ίσως ε, καταλαβαίνετε γιατί περίμενα την ε, Κομισιόν. Καταρχήν είναι αυτή η σωστή σειρά. Αλλά από την άλλη θεωρώ ότι είναι σημαντικό να οπτικοποιούνται τα πράγματα για να τα κατανοήσει κανείς καλύτερα. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό, πολύ καλή αυτή η δουλειά. Την επόμενη εβδομάδα είναι... Αυτή είναι η συνάντηση αυτή, τελευταία ήταν τον Ιανουάριο και πρόκειται για ένα θέμα που θα βελτιώσει σημαντικά την κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, και των ανθρώπων με αναπηρία, αν σκεφτεί κανεί ότι κάποτε θα υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα στην Ευρώπη μαζί με την ε, ψηφιοποίηση και το shared economy ε, θα βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες για αυτούς τους ανθρώπους και βεβαίως είναι σημαντικό να έχουμε πράγματι τα δεδομένα στη διάθεσή μας. Έχουμε ήδη συζητήσει και έχουμε πει τις απόψεις μας. Θα ήθελα να θέσω τι εξής ερωτήσεις. Πρώτον, πώς ε, ε, όλες οι χώρες μεν συμμετέχουν, αλλά σε ορισμένε χώρες είναι δύσκολο να βγάλουν τα δεδομένα, δώσουν τα δεδομένα. Στη Γερμανία, ε, όπως ξέρετε, δεν είναι ρόδινα τα πράγματα με τους σιδηροδρόμους και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντλήσουμε τα στοιχεία της πληροφορίας. Αφενός πρόκειται για τα συμφέροντα των μονοπωλίων, τα οποία πράγματι υφίστανται και είναι δύσκολο να σπάσουν. Ε, και κάτι άλλο. Ξέρω ότι γίνεται στο Αμβούργο καλύτερα από τις άλλες γερμανικές πόλεις. Ο γιος μου που σπουδάζει εκεί λέει ότι δεν, δεν χρειάζεται αυτοκίνητο ότι έχει μια πληθώρα πληροφοριών εάν βάλει στο σύστημα το μέρος το οποίο βρίσκεται και τον ε, μέρος το οποίο θέλει να μεταβεί. Και κάτι τέτοιο πραγματικά θα ήταν ιδεώδες για ολόκληρη την Ευρώπη. Το ερώτημα άρα είναι πού βρίσκονται τα εμπόδια και πώς μπορούμε εμείς οι βουλευτές να συμβάλλουμε ούτως ώστε να ασκήσουμε πίεση στο επίπεδο των χωρών μελών, γιατί πραγματικά ε, θα ήταν προς συμφέρον μας και είναι καλό και για το περιβάλλον και για... θα είναι ε, μεγαλύτερη οικονομία. Ευχαριστώ. Η ασυμβατότητα και η ασυνέπεια των δεδομένων και η ελλειπής διαλειτουργικότητα των ε, φόρματων δεδομένων αποτελούν πρόβλημα για μια ευρωπαϊκή ανταλλαγή πληροφοριών και παροχή πληροφοριών για τις πολυτροπικές μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ως εισηγητής για την έκθεση αυτή χαίρομαι που θέλουμε να καταλήξουμε τελικά σε ένα σύστημα ευρωπαϊκό για την ε, ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών και την παροχή των πληροφοριών αυτών. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα και βεβαίω να είναι τα δεδομένα αυτά και ε, ε, επίκαιρα και έγκαιρα. Η ανταλλαγή θα πρέπει να μπορεί να γίνει. Υπάρχουν πολύ πιο ακριβή δεδομένα για αλλαγές ε, των δρομολογίων κτλ. Άκουσα κάποια σχόλια σχετικά και σημαντικό ήταν πάντα για μας να έχουμε ανοιχτούς κόμβους και καλό ήταν η να ληφθεί αυτό υπόψη στην επεξεργασία της κατεξουδότησης πράξης. Και ένα ερώτημα. Έχουμε ένα σημαντικό σημείο για την προσβασιμότητα των δεδομένων σε ό,τι αφορά την, ε, την ε, κινητικότητα των ε, ατόμων με αναπηρία. Πάντα το θεωρούσαμε σημαντικό αυτό και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν θα συντάξετε την κατεξουδότηση πράξη. Ευχαριστώ. Ο Γιάννης έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ήμουν σκιώδης εισηγητής για αυτή την έκθεση. Νομίζω είναι σημαντικό να συζητήσουμε την ανάγκη για τη δημιουργία ενό φόρουμ όπου οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε διάφορα Ήδη εταιριών που ασχολούνται με αυτό το θέμα, εταιρείε μεταφορών που ενδιαφέρονται για αυτή την πρωτοβουλία, για αυτά τα βήματα. Οπότε θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τέτοιο φόρουμ. Ευχαριστώ. Έγραψα και εγώ το δικό μου όνομα στην ε, λίστα για το σύστημα που υπάρχει στο Αμβούργο, που υπάρχει και στο Βερολίνο και νομίζω ότι εκεί υπάρχουν καλά δεδομένα. Ε, βάζω τα δεδομένα εγώ στο σύστημα από τη σημείο που είμαι και έχω όλα τα δεδομένα για το ποια είναι τα λεωφορεία που περνούν από εκεί, τα τρένα που περνούν από εκεί κτλ. Στη Γερμανία έχουμε καλό σύστημα στους γερμανικούς ε, σιδηροδρόμους. σε όλη την, ε, μπορώ να, πάρω τα, να βρω ποιες είναι οι συνδέσεις των τρένων, αλλά θα ήθελα να δω το το σύστημα πώς λειτουργεί ας πούμε από το Ταλίν σε μια άλλη πόλη. Δεν υπάρχουν εκεί δεδομένα. Μπαίνω όμως στο ίντερνετ και ψάχνω να βρω μια σύνδεση από το Ταλίν με άλλη πόλη και τη βρίσκω. Βεβαίως τα διάφορα συστήματα πρέπει να συνδυαστούν. Υπάρχει και το τρίτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους που χρονολογείται από το 2006-2007 και τα είχαμε αποφασίσει όλα τότε και οι σιδηρόδρομοι ήταν το, ε, είναι οι τελευταίες εθνικιστικές αρχές ας πούμε που αρνούνται να μπουν στο σύστημα τα, δεδομένα υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και, τα, και το γνωρίζουν ότι αν δεν μπουν στο σύστημα αυτό τότε θα το κάνουμε εμείς υποχρεωτικά και τέλος Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται λοιπόν. Εσείς όμως τι πίεση έχετε ασκήσει και τι δυνατότητες έχουν οι ε, σιδηρόδρομοι που εδώ και χρόνια αρνούνται να ενταχθούν στο σύστημα για τον οποιοδήποτε λόγο Κανένα επιχειρηματία δεν θα έκανε τίποτα τέτοιο, γιατί θα ήταν προ όφελό του να μπει στο σύστημα. Δεν το καταλαβαίνω λοιπόν εγώ. Εσεί πώ μπορείτε λοιπόν να ασκήσετε τέτοιες, τέτοια πίεση ώστε να έχουμε τι πληροφορίε. Και δεν μιλούμε μόνο για τι πληροφορίε, για να μην μπω σε, σε πληροφορίε για τι ε, τιμέ και για τα εισιτήρια κτλ. Για, για τι αερομεταφορέ υπάρχουν αυτά. Μια αντιγραφή απλώ χρειάζεται. Αλλά έχουν καταλάβει εν μεταξύ οι αρχέ των σιδηροδρόμων τι θέλουμε να κάνουμε. Και εσεί έχετε ασκήσει πίεση, γιατί εμεί θα προχωρήσουμε ούτω ή άλλω. Ο Ντομινίκ έχει το λόγο. Εγώ είμαι ιδιαίτερο ε, ικανοποιημένος που προχωράμε στο θέμα αυτό. Είναι αλήθεια ότι υπήρξαν πολλές δυσκολίε όπω είπε η εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Έχω δύο ερωτήματα να θέσω που αφαιρούν την, ε, το δυναμισμό του συστήματος από τη μία και τη δυνατότητα να εξελιχθεί το σύστημα. Κατά πόσο η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι ευκταίο να οριστούν κάποιοι κανόνες με όλες τις δυσκολίες που θα ανακύψουν. Γιατί οι δυσκολίες με τους κανόνες είναι ότι μετά από τρία χρόνια μπορεί να ξεπεραστούν. Έχει η Κομισιόν κάποια ιδέα πώς, μπορεί, πώς μπορούν να διατυπωθούν αυτοί οι κανόνες και δεύτερον, είναι σημαντικό να υπάρξει ένα συγκεντρωτικό σύστημα, ούτως ώστε το σύνολο αυτών των δεδομένων να μπορούν να μεταφερθούν σε αυτό το κεντρικό σύστημα. Ή μήπως θα ήταν προτιμότερο να υπήρξαν διασυνδέσεις σε πλατφόρμες ε, που θα παρέχουν αυτές τις πληροφορίες. Ε, άρα το θέμα είναι κατά πόσο είναι φταίο να υπάρξει ένα άκαμπτο σύστημα, κεντρικό σύστημα ή μήπως θα ήταν καλύτερο να προτιμήσουμε ένα σύστημα όπως αυτό που έχουμε για τις και κυκλοφορίες όπου θα υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης και όπου θα προτιμήσουμε να υπάρξει δυνατότητα διασύνδεση, θα την προτιμήσουμε από μια κεντρική διαχείριση των δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η Κάρεν Μαντέλη. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα εντάχει να ρωτήσω την Επιτροπή το εξής. Καταρχήν, πώς έχετε συμπεριλάβει ακριβώς τα εμπόδια ε, προσβασιμότητας ε, στα διάφορα φορμάτ των πληροφοριών ε, που αφορούν τις πολυτροπικές μεταφορές. Δεύτερον, υπάρχει κάτι στις πληροφορίες σας που να μας αφορά άμεσα όσον αφορά τις, τη διασύνδεση πληροφορίες που αφορούν την ενεργειακή κατανάλωση, τις κλιματικές επιπτώσεις και λοιπά των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Ευχαριστούμε. Τώρα ο Παπαλ Λίτσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την πρόσωπο τη Κομισιόν. Ήθελα και εγώ να προσεγγίσω το θέμα αυτό από με μια, από μια παρόμοια οπτική όπω η δική σα. Νομίζω ότι έχουμε λάβει κάποιε πληροφορίε για το τι συμβαίνει. Τα α, πρότυπα βασικά είναι το πρόβλημα. Αλλά όπω είπατε, οι πληροφορίε είναι διαθέσιμε. Το ερώτημα είναι να υπάρξει αμοιβαία αποδοχή και αμοιβαία εναρμόνιση. Κάτι που δεν είναι βεβαίως εύκολο και είναι και αρκετά ε, κοστοβόρο. Αλλά αυτό δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Το πρόβλημα, ο πυρήνος του προβλήματος είναι ότι οι εταιρείε, οι σιδηροδρομικές και όχι μόνο αυτές, δεν θέλουν καν να ασχοληθούν. Όταν ήμουν ασκιώδης για τον ε, κύριο Κόχ έκανα ε, πολλές επαφές με διάφορους εκπροσώπους εταιριών κτλ. Και, και βλέπετε ότι για αυτούς αυτό το ζήτημα τα πρότυπα δηλαδή είναι το τελευταίο εργαλείο που θέλουν να χρησιμοποιήσουν για να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και ενώ η κατεξοδότηση πράξη μπορεί βεβαίω να συμβάλλει με προθεσμία τελική το 2019, που εντάξει μπορεί να είναι καλό, Νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πιέσουμε και με τόσο ό,τι αφορά την, το ολοκληρωμένο σύστημα για την έκδοση εισιτηρίων. Ε, η Κομισιόν ίσως θα πρέπει να ε, μπλακεί πιο αποτελεσματικά σε αυτό, γιατί αυτό είναι αυτό περί του οποίου μιλούμε. Δεν θέλουμε να είναι απλώ διαθέσιμε πληροφορίε. θέλουμε να είναι χρήσιμε, να μπορούν να διευκολύνουν τους καταναλωτές, τους πελάτες. Αυτό είναι το θέμα. Στα πλαίσια βεβαίως τη συνολικής απελευθέρωση. Το ίδιο κάναμε και με το τέταρτο πακέτο για τους υδροδρόμους. Το ίδιο θέμα αντιμετωπίζουμε. Και το Κοινοβούλιο πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό. Δεν έχω κάποια ερώτηση να θέσω. Σίγουρα είναι καλή η προσέγγιση της Κομισιόν, αλλά θα ήθελα κι εγώ να συμφωνήσω με τα όσα είπε η συγκήτρια. Τι μπορούμε να κάνουμε για να διευκολύνουμε περισσότερο όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Πολλά λοιπόν τα ερωτήματα προς την Κομισιόν και περιμένουμε εναγωνίως τις απαντήσεις σας. Thank ευχαριστώ. Με χαρά βλέπω ότι το θέμα σας ενδιαφέρει. αρχίσαμε πρώτες παρατηρήσεις. Ναι, έχετε δίκιο. Έχουμε αυτό το πακέτο για τα δικαιώματα των ποιοτών. Άλλη μια νομοθεσία δηλαδή προσπαθήσαμε να προωθήσουμε. σιδηρόδρομοι. Ο κ. Νίλσεν νομίζω είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια κατάσταση που θα ικανοποιεί τους πάντες. Win-win. Δίκιο έχετε. Μην ξεχνάμε όμω ότι ταυτόχρονα και οι σιδηρόδρομοι παρέχουν πληροφορίες. Και αυτοί λοιπόν επιθυμούν να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις δημόσιες μεταφορές. Τα πράγματα λοιπόν μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση πάνε. Επειδή έχετε περισσότερους επιβάτες, περισσότερους πελάτες, αλλά ταυτόχρονα μπορείτε να παράσχετε κάτι επιπλέον, κάτι συμπληρωματικό πέραν της έκδοσης του εισιτηρίου. Να πούμε λοιπόν όλοι ότι αυτό που θέλουμε είναι να καλύψουμε αυτές τις μετακινήσεις από ένα συγκεκριμένο σημείο σε ένα άλλο σημείο με τρόπο ολοκληρωμένο. Μειωμένη κινητικότητα. Έχετε δίκιο. Αυτό πρέπει να αποτελεί τη βάση ενός πολύτροπου ταξιδιού. Έχουμε να κάνουμε με θέματα δικαιωμάτων, πρόσβασης σε συνδρομικούς σταθμούς, αερολιμένες, πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες κλπ. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε όσο γίνεται όλες τις καταστάσεις. Αλλά και πάλι εδώ μιλάμε για την παροχή δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν όταν θα είναι διαθέσιμα τα δεδομένα, όταν δηλαδή ο πάροχος των υπηρεσιών θα είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσει. Ερώτηση του κυρίου Ρικέ. Όλα να γίνονται κεντρικά. Σε επίπεδο μέχρι τελευταίες λεπτομέρειες είναι να έχουμε κάτι πιο ευέλικτο. Κοιτάξτε την ε, οδηγία ITS. Θέλαμε όλοι αρχικά να υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο είναι ευέλικτο. Αυτή ήταν η εντολή που μας δώσατε. Προσπαθήσαμε βεβαίως να πάμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όχι χωρίς παραπομπή σε προδιαγραφές. Το αντίθετο. Θέλουμε λοιπόν στη φάση εφαρμογή να καλύψουμε όσε περισσότερε καταστάσει ε, γίνεται, Χωρί να έχουμε αυτέ τι επιλογέ που έχουμε στην διαφάνεια. Εθνικά σημεία πρόσβαση κλπ. Αυτή την εμπειρία είχαν και οι Ολλανδοί συνάδελφοι. Έχουμε ένα χώρο αποθήκευση των δεδομένων ή μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα άλλο μοντέλο, μοντέλο που ήδη εφαρμόζουν ε, διάφορε άλλε χώρε μέλη. Μπορούμε να το δούμε αυτό το χώρο προσβεδομένο σε ένα είδο βιβλιοθήκη. Δηλαδή Πάω πάρω το βιβλίο, βλέπω στο κατάλογο ότι είναι θέσιμο το βιβλίο, σε συγκεκριμένη θέση και ξέρω ακριβώ ποιοι είναι οι όροι χρήση του βιβλίου αυτού. Στη δική μα περίπτωση τα δεδομένα. Νομίζω ότι απάντησα για τις προδιαγραφές. θα μπορούσαμε να είχαμε παρακάμψει όλε τι διαδικασίε τυποποίηση και να πούμε ότι εντάξει αφού ο συνδρόμο έχει δικιά τις, τις δικές η αεροπλογία τι δικέ τη κτλ. Δεν τι χρειαζόμαστε. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα ήταν χρήσιμο και εφαρμόσιμο. Οπότε καμιά φορά πρέπει να δούμε και τι θέλουμε. Δηλαδή να έχουμε ένα τέλειο σύστημα το οποίο αν ποτέ υλοποιηθεί θα γίνει σε 15 χρόνια ή θέλουμε σιγά σιγά να προοδεύουμε και να προχωράμε με μικρά βήματα. Ας είμαστε λοιπόν ρεαλιστές. Τα δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τον σιδηρόδρομο θα συνεχίζουν να παρέχονται σε αυτό το πλαίσιο όπως ακριβώς ζητά και η οδηγία TSI. Η διαφορά είναι όμως ότι όταν ένας πάροχος να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα ξέρουν, ξέρουν ότι υπάρχουν δεδομένα τα οποία είναι διαθέσιμα υπό ποια μορφή κλπ και είναι πολύ πιο εύκολο να μεταφερθούν και να μεταφραστούν κατά κάποιο τρόπο αυτά τα δεδομένα προς τους χρήστες. Να σας διακόψω, λέει ο Πρόεδρος. Το Voodoo, αυτή η εφαρμογή. Έχω εκατοντάδες πληροφορίες για τις πτήσεις στο Βερολίνο. Με μία εφαρμογή. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν για τους σιδηρόδρομους να έχουμε μία εφαρμογή που θα μας δίνει όλες αυτές τις πληροφορίες γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά λοιπόν. Γιατί, γιατί. Απάντηση. Εντάξει, θα έρθω και σε αυτό. Αλλά μιλάμε για μια εφαρμογή και μόνο δεν είμαι βέβαιη. Ίσως λόγω μητρότητας να με ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες που αφορούν τα μικρά παιδιά με το καρότσι και τα λοιπά. Τι πληροφορίες θέλω εγώ. Αλλά Εγώ σας έλεγα τι προσπαθούμε να αναπτύξουμε ως τεχνικό θέμα, θέμα διακυβέρνησης και κυρίως θέλουμε να δούμε κατά πόσο ας πούμε ο συγκεκριμένος πάροχος εδρομικών υπηρεσιών διαθέτει τα στοιχεία του και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ας πούμε, στο σιδηρόδρομο είναι πιο ορατοί, είναι πιο προσβάσιμοι για τους χρήστες. Ο κύριος Νέφης νομίζω είπε Τι γίνεται με τους φορείς των μεταφορών, συζητάτε με αυτούς. Ναι, εντάξει, συζητάμε. Αλλά αυτή η νομοθεσία θα εφαρμοστεί όχι με την προπόθεση ότι θα διαθέσουμε αυτά τα στοιχεία, είναι υποχρεωτικό, θα πρέπει να εφαρμοστεί ούτω ή άλλω. Οπότε λοιπόν, αφού υιοθετηθεί η νομοθεσία αυτή, εφαρμόζεται. Αν λοιπόν ένα μεταφορέα ή ένα πάροχο μεταφορών τέλο πάντων έχει τα δεδομένα αυτά τα ψηφιακά, τότε θα πρέπει να εφαρμόσει τις διάφορες διατάξεις που περιλαμβάνει η κατεξουσιοδότηση νομοθεσία. Να έχουμε λοιπόν μια πιο νομοτεχνική προσέγγιση λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα. Δεν ξέρω. Προσπαθούμε να δώσουμε κάποια ευελιξία ώστε να επιτρέψουμε τα διάφορα αυτά μοντέλα να εφαρμοστούν στις διάφορες χώρες, αλλά αφήνοντας και περιθώριο την εμφάνιση και δημιουργία νέων υπηρεσιών με τρόπο έτσι ρεαλιστικό. Κάτι άλλο ακόμα. Η εμπλοκή των διαφορών φορέων μεταφορών. Συζητήσαμε με τους εκπροσώπους του σιδηροδρόμου, τους παρουσιάσαμε τι θέλουμε να κάνουμε στη Διευθύνουσα Επιτροπή του ΤΑΠ. Συναντήκαμε λοιπόν επανειλημμένως μαζί τους, με τους ιεροδρομικούς και μια συνάδελφο σήμερα συναντιέται μάλιστα με τους εκπροσώπους του τομέα των δημοσίων μεταφορών. Αν δούμε λοιπόν όλη αυτή την αλυσίδα, στις δημόσιες μεταφορές έχουμε χαμηλότερη παρουσία των ψηφιακών δεδομένων. Οπότε θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως ευκαιρία για την προώθηση της χρήσης των δημοσίων μεταφορών. Αυτά. Και λέω να κλείσω με την έκδοση των εισιτηρίων. Δεν γίνεται ότι, μάλλον δεν ισχύει ότι δεν γίνεται τίποτα εκεί. Έχουμε την ευκαιρία του ορίζοντα 2020 Έχουμε τα ΣΕΦ ως ε, ευκαιρίες ή δυνατότητες χρηματοδότησης. Ανακύπτουν προγράμματα, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό σημείο. Έχουμε και το τέταρτο πακέτο για το σιδηρόδρομο. Εδώ πέρα χαράζουμε μία κατεύθυνση. Εγώ ίδια δεν παρακολούθησα από κοντά τις διαπραγματεύσεις, αλλά υπάρχει ένα εργαλείο πίεσης εδώ. Μπορούμε λοιπόν να προωθήσουμε και τα δύο παράλληλα και κάποια στιγμή στο μέλλον, επειδή θεωρώ ότι υπάρχει και κάποια ρήτρα θεώρηση εδώ, έτσι, και χρονικά δεν είναι και τόσο μακριά αυτό. Να δούμε λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε, να σημειώσουμε πρόοδο και στο συγκεκριμένο πλαίσιο εδώ θέλουμε να έχουμε εθνικά σημεία πρόσβασης τα οποία θα ήδη έχουν υλοποιηθεί και θα λειτουργούν το 19. Το 19, ξέρετε, μία μόνο τρία χρόνια, έτσι. Δρόμος. Ευχαριστώ. Γεζίνα. Ναι, δεν έχω να πω και πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενημερωνόμαστε για τις περαιτέρω προόδους. Βεβαίως, συμμερίζομαι κάπως την ανησυχία, την ανυπομονησία του Προέδρου ε, γιατί πραγματικά αν επιταχυνθούν τα πράγματα του σιδηροδρόμου θα ήταν τεράστιο βήμα προς τα μπρο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είμαστε στον καλό δρόμο και βεβαίω τόσο η Κομισιόν όσο και οι χώρε μέλη θα πρέπει να ασκήσουν πίεση και θα πρέπει στις διμερείς συζητήσει με τι χώρε μέλη να δούμε κατά πόσο οι διαφερόμενοι, οι ενεχόμενοι θα μπορούν ε, να ε, παρατηρηθούν προς τα μπρος. Ευχαριστώ. Επειδή είμαστε κάτω από πίεση χρόνου, θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας ε, διάταξης που αφορά το κανονισμό της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού αναφορικά με την εφαρμογή ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών. Στον εκπρόσωπο της Επιτροπής θα δώσω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας παρουσιάσω σήμερα το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού και για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των επιχειρήσεων ε, οδικών μεταφορών. 28 Ιανουαρίου ψηφίστηκε το κείμενο και έχει έρθει στο Κοινοβούλιο για να το μελετήσετε. Πριν ε, πάω πολύ γρήγορα στο βασικό σημείο του εφαρμοστικού κανονισμού, δύο λόγια που σίγουρα θα ξέρετε. Το σύστημα αυτό ισχύει. Υπάρχει ήδη, είναι ο κανονισμός του 2010 που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις του συστήματος που σημαίνει ότι το σχέδιο εφαρμοστικού κανονισμού είναι απλώς ε, μια αναβάθμιση του μηχανισμού, αλλά ε, σημαντική αναβάθμιση. Ε, δεν χρειάζεται να σας θυμίσω την σημασία του συστήματος αυτού που είναι πολύ σημαντικό για την εφαρμογή. Ο μηχανισμός λοιπόν επιτρέπει την διασύνδεση των εθνικών ε, μητρώων για, τους, ε, για τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών. Πολύ σημαντικό εργαλείο λοιπόν για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Σίγουρα θα γνωρίζετε ότι πολλά κράτη-μέλη δεν συμμορφώθηκαν με την προθεσμία για τη διασύνδεση των εθνικών τους μητρών με το ΕΡΟΥ ε, με την 31η Δεκεμβρίου του 2012 δηλαδή, ο ε, λόγος για, τον οποίο, λόγος η Κομισιόν ξεκίνησε με διάφορες διαδικασίες επεραβάση το 2015 που ήταν ε, αρκετά επιτυχίες. Τώρα έχουμε 23 κρατημέλη τα οποία έχουν συνδέσει τα εθνικά τους μητρώα με το ευρωπαϊκό. Ε, επίσης, η διαδικασία αυτή ε, συνεχίζεται. Κάποια, τέσσερα κρατημέλη έχουν ε, κάποια δυσκολία να κατανοήσουν ε, ποια είναι η σημασία του να συνδέσουν το εθνικό του μητρό με το ευρωπαϊκό και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο η Κομισιόν έχει ξαναξεκινήσει διαδικασία επί παραβάση για αυτά τα τέσσερα κρατημέλη και τα έχει παραπέμψει στο δικαστήριο. Κάποια σχόλια τώρα για το σχέδιο του εφαρμοστικού κανονισμού. Υπάρχουν τέσσερα βασικά καινοτόμα στοιχεία για το σύστημα αυτό. Το πρώτο είναι μια τροποποίηση το, της δυνατότητας ανταλλαγής μηνυμάτων με σκοπό να βελτιωθεί η απόδοση της έρευνας και των πληροφοριών που λαμβάνονται. Δεύτερο καινοτόμο στοιχείο είναι μια νέα λειτουργία που υπάρχει μέσω του νέου μηχανισμού ε, θα είναι δυνατό να ανταλλάσσονται πληροφορίες για την άδεια του, ε, της επιχείρησης και για την ισχύ αυτής της άδειας. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, οι ε, ελεγκτές ε, των ε, τροχιών σημάτων να έχουν το ρόλο που τους αρμόζει, γιατί προς το παρόν έχουμε τον έλεγχο μόνο των αδειών, αλλά θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα αρκετά σημαντικό βήμα. Και τέταρτον, ε, τέταρτο, τέταρτη κοινοτομία, υπάρχει μια προσαρμογή του Ευρωπαϊκού Μητρώου στην ανταλλαγή πληροφοριών για σοβαρές και πολύ σοβαρές πληροφορίες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί η Κομισιόν ε, θα υιοθετήσει μετά τη θετική γνωμοδότηση του, του, του Κοινοβουλίου τον κανονισμό για τις σοβαρές παραβάσεις. Ε, οπότε νομίζω ότι θα έχουμε ένα επαρκές ε, έτσι, εργαλείο, ένα επαρκή ε, ευρωπαϊκό μηχανισμό και μαζί με τον κανονισμό που θα περιμένουμε να εγκριθεί για τις ε, σοβαρές παραβάσεις, μια κοινή γλώσσα για την ανταλλαγή πληροφοριών για τέτοιου είδους παραβάσεις. αυτά λοιπόν, αυτό είναι το πνεύμα του σχεδίου κανονισμού. Αυτή είναι οι κανόνες που το διέπουν και για να κλείσω Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει στεναρά αυτό το σχέδιο εφαρμοστικού κανονισμού. Αυτά, Πρόεδρε, μένα ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Θέλει κάποιο το λόγο. Κυρία Νίλσεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή αυτή. Χθες ε, συζητήσαμε μια γνωμοδότηση σε σχέση με τον δίκαιο ανταγωνισμό και το social dumping, το κοινωνικό dumping. Και νομίζω ότι υπήρξε μια ευρεία συνένεση για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου του κοινωνικού dumping. Χρειαζόμαστε λοιπόν την ύπαρξη κανόνων στις χώρες μέλη, την ύπαρξη αποτελεσματικών ελέγχων και ακούσαμε μια πρόταση για την εξαίρεση των μικρών επιχειρήσεων που διαθέτουν μόνο ή ένα-δύο φορτηγά. Θα ήθελα να πείτε την απόψή σας γι' αυτό. Δηλαδή για την εξαίρεση επιχειρήσεων που δεν έχουν σημαντικό εξοπλισμό. Επίσης, για την περίπτωση όπου ένα ελεκτής ας πούμε σταματήσει ένα φορτηγό μια τελίκα που έρχεται από την Τσεχία θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα τα εθνικά της ε, Τσεχίας όσον αφορά και τον οδηγό αλλά και το όχημα. Είναι σημαντικό να υπάρχει λοιπόν δυνατότητα πρόσβαση σε όλε τι βάσει δεδομένων, αν θέλουμε η έλεγχη να είναι αποτελεσματική. Αυτά από μένα, αυτέ οι ερωτήσει. Ευχαριστώ κυρία Καρυμαντελή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση της Κομισιόν. Να μου πείτε, αυτές οι ηλεκτρονικές ανταλλαγές ανταποκρίνονται στις απαιτήσει διαλειτουργικότητας με τα συμβατικά συστήματα. Μπορείτε να μας το επιδέσετε αυτό σήμερα Κομισιόν. Να, επειδή δεν υπάρχουν άλλες ε, παρεμβάσεις, θα δώσω και πάλι το λόγο στην ε, Επιτροπή. Θα επαναλάβω την ερώτηση Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο αυτή η ηλεκτρονική ανταλλαγή ανταποκρίνεται στις απαιτήσει της ε, πολυτροπικότητας με το συμβατικό σύστημα. Διαλειτουργικότητα, συγγνώμη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Όσον αφορά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχει προβλεφθεί ένας εφαρμοστικός κανονισμός όσον αφορά μια εξαίρεση. Γιατί θα πρέπει η αστυνομία να είναι σε θέση να ελέγχει επιχειρήσεις είτε είναι μεγάλες είτε είναι μικρές. Δεν προβλέπεται λοιπόν εξαίρεση Ωστόσο, η προσπάθεια έρευνας εναπόκειται στις χώρες μέλη. Όσον αφορά την διαλειτουργικότητα, δεν υπάρχει πραγματικά διαλειτουργικότητα. Το σύστημα ΕΡΟΥ, το Ευρωπαϊκού Μητρώου για τις Επιχειρήσεις Ειδικών Μεταφορών, βασίζεται σε ένα σύστημα ανταλλαγών και δουλεύει αυτούσια Επίσης έχουμε προβλέψει άλλα συστήματα βάσης δεδομένων, τα οποία θα μοιράζονται περισσότεροι, τα οποία βασίζονται στην ε, ίδια τεχνολογία και θα αφορά ανταλλαγές πληροφοριών για αδειοδοτήσεις και για τους, ε, ε, τις των οχημάτων. Τα ταχόμετρα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τώρα <laughs> τελειώσαμε τόσο γρήγορα που έχουμε ένα ολόκληρο τέταρτο στη διάθεσή μας. Στις 11 ακριβώς θα έρθει η Επίτροπος ε, κυρία Πιενκόφσκα και Task Force για τον τουρισμό. Και πάλι έχουμε ένα τέταρτο διάλειμμα. I think we can start. Μπορούμε. να ξεκινήσουμε νομίζω. Hm? wir kommen nun zu unserer Sitzung der Πάμε λοιπόν στην ειδική ομάδα για τον τουρισμό και Έχουμε τον πρόεδρο της ειδική ομάδας για τον τουρισμό και θα ήθελα από κοινού να καλωσορίσουμε την Επίτροπο Ελσβιέτα Μπιενκόφσκα. Είναι πρώτη φορά που έρχεται εδώ για να μας μιλήσει. Τελευταία φορά που είχαμε επίτροπο εδώ παρόντα για τον τουρισμό ήταν ο Επίτροπος Ταγιάννη το 2013. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ κυρία Επίτροπε και βεβαίως με χαρά θα ακούσουμε την παρουσίασή σας. Μετά θα δώσουμε το λόγο στην, ε, στον πρόεδρο, τον Ethan Way, για την ε, ειδική ομάδα για τον τουρισμό, για να μας ε, κάνει και αυτός τη δική του παρέμβαση και μετά θα κάνουμε τη συζήτηση. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Thank you very much, Chairman, members. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε βουλευτές. Έχει πέρασει πολλής χρόνος που η Επιτροπή αυτή έχει να συζητήσει θέματα τουρισμού με επίτροπο. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν που με προσκαλέσατε για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά την κυρία Ντεμόντε για την πολύ καλή έκθεση για τις νέες προκλήσεις και έννοιες στην πρόθεση του τουρισμού στην Ευρώπη που θετήθηκε πέρσι λέχει θαυμάσιες ιδέες και συστάσεις που εξετάζουμε και τις οποίες αναφέρω και στη συνέχεια. Στην Επιτροπή, όπως ξέρετε, δεν έχουμε μεγάλη ποικιλία εργαλείων για τον τουρισμό. Θέλουμε όμως να είμαστε πιο ενεργοί, ξεκινώντας από τώρα. Έχουμε την τουριστική στρατηγική του 10 βάσει τις οποίες θα θέλαμε να είμαστε έτσι πιο ενεργοί σε κάποια σημεία που αφορούν τον τουρισμό. Να επιθυμίσω κάποια πράγματα, ξέρετε καλύτερα από μένα. Ο τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή οικονομία, αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των ΑΕΠ μας. Το 2014, άμεσα ή έμεσα, υποστήριξε 24 εκατομμύρια θέσεων εργασίας, 10% δηλαδή του συνολικού ΑΕΠ της Ένωσης. Αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό, ο σημαντικός ρόλος της βιομηχανίας μας, γιατί έτσι εγώ την αντιλαμβάνομαι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ευημερία και την ανάκαμψη. Και παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα βέβαια. Ο τουρισμός και σχετίζεται με άλλες βιομηχανίες, μεταφορές, λιανικό εμπόριο, πολλές άλλες δηλαδή δημιουργικές βιομηχανίες. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε δυσκολίες η ευρωπαϊκή οικονομία, όμως ο τουρισμός και οι δημιουργικές βιομηχανίες ήταν οι δύο τομείς, οι δύο κλάδοι που αποδείχτηκαν πιο ανθεκτικοί στην κρίση. Όσο βελτιώνεται λοιπόν η οικονομία, περιμένουμε να αυξηθεί και ο τουρισμός. Ξέρουμε ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Θα απαριθμίσω κάποιες από αυτές. Κάποιες μοιάζουν με αυτές που αντιμετωπίζουν οι άλλοι κλάδοι. Κάποιες είναι ιδιαίτερες στο τουρισμό. Καταρχάς η ψηφιοποίηση και η εμφάνιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, η συνεργατική οικονομία και η αλλαγή της στάσης των καταναλωτών. Τα παραδοσιακά μοντέλα τουρισμού νομίζω γίνονται παροχημένα. Οι καταναλωτές αναζητούν νέο είδος διακοπών στα μέτρα τους άμεσα διαθέσιμα και η βιομηχανία βέβαια πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό. Μετά έχουμε αυξημένο ανταγωνισμό από νέου προορισμού, αυξάνονται οι αριθμοί των τουρισμών, αλλά το μερίδιο αγορά μειώνεται. Να φερθώ σε δύο στοιχεία συγκεκριμένα. Το 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήχε το 50% τη παγκοσμία αγορά. Σήμερα είμαστε κάτω από το 40% και προβλέπεται περαιτέρω μείωση στο 31% το 2030. Τρίτον, η πρόκληση όσον αφορά τι αξιότητε η διασφάλιση δεξιοτήτων και επιχειρηματικών και ψηφιακών ώστε να αποφεληθεί ο κλάδος. Επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το 99% των επιχειρήσεων σε αυτό το τομέα είναι μικρομεσαίες. Οπότε βλέπετε θα μπορούσα να σας είχα παριθμίσει και άλλες προκλήσεις που αναφέρονται στο πρόσφατο ψηφισμά σας. Αλλά νομίζω ότι εδώ έχουμε μια ευκαιρία την οποία θα πρέπει να δράξουμε η πρώτη ας πούμε πρόκληση, συνεργατική οικονομία και ψηφιοποίηση. Σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ευφυή και βιώσιμα προϊόντα τουριστικά. Αυτό ψάχνουν και οι τουρίστε σήμερα. Με μια καινοτόμο προσέγγιση νομίζω ότι οι πιθανότητε είναι πολλέ. και αυτό ήδη σημαίνει τώρα σε πολλού τομεί τη βιομηχανία μα, Δεύτερη πρόκληση α πούμε, η, δεύτερη, η αύξηση του ανταγωνισμού από τρίτε χώρε. και πάλι αυτό θα μπορούσε κανεί να πει ότι αποτελεί μια ευκαιρία για να προσελκύσουμε τουρίστε εκτό Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τι προσπάθειές μα για να κάνουμε την Ευρώπη πιο παρούσα, πιο ορατή ως τουριστικό στόχο. Μετά, οι δεξιότητε. Και πάλι, αυτό είναι μια ευκαιρία για του νέου με νέε δεξιότητες να μπουν στην αγορά. Ανταποκρινούμε λοιπόν στι προκλήσει αυτέ σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε προσαρμογή των επιχειρήσεων. Σημαίνει όμω ότι και αυτέ οι επιχειρήσει θα πρέπει να συνεργαστούν. Θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία μαζί με άλλους τομείς όπως η μόδα, οι μεταφορές κτλ. Και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κομμάτι των μελλοντικών μας δραστηριοτήτων στην Κομισιόν, ώστε να προετοιμάσουμε κάποιες κατευθύντες γραμμές και ένα σχέδιο δράσης, ώστε να υπάρχει η σύνδεση μεταξύ τουρισμού και τομέων ή κλάδων όπως μεταφορές, μόδα κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να διαθέτουν οι μελλοντικοί εργαζόμενοι τις κατάλληλες δεξιότητες. Επίσης, οι οργανώσεις του κλάδου θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο εδώ. Ε, πρόσφατα είχαμε ένα μανιφέστο τουριστικό που δημοσιεύτηκε ώστε να προσαρμοστεί και να καλύψει το κοινό βιομηχανία, να αποφυληθούμε από τις προσπάθειες ψηφιοποίησης στις διάφορες χώρες και να χρησιμοποιηθούν σωστά οι πλατφόρμες του ίντερνετ. Πρέπει επίσης να προωθήσουμε τις δεξιότητες μέσω στάζ που θα πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να ε, έχουμε καλύτερη διασύνδεση με τις τοπικές και εθνικές αρχές ώστε να βελτιωθεί η συμμετοχή των τοπικών παραγόντων στον κλάδο του τουρισμού. Θα πρέπει βέβαια να υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες για να πετύχει η βιομηχανία μας. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε φραγμούς, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να προωθήσουμε την Ευρώπη να συνεργαστούμε. Στην Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή εμείς θέλουμε να διαδραματίσουμε πλήρως τον ρόλο μας εδώ και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε μια συντονισμένη προσέγγιση. Στοχεύουμε λοιπόν σε διάφορους τομείς όπου θεωρούμε ότι υπάρχει περισσότερη αξία. Να παρθυμίσουμε λοιπόν κάποια μέτρα τα οποία λαμβάνουμε και τα οποία θεωρούμε θα βοηθήσουν τον τουριστικού κλάδο να ανταποκριθεί. Καταρχά, η δημιουργία ευκαιριών. Κύριο σημείο εδώ είναι το να έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση ο τουριστικός κλάδος, ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για εξυγχρονισμό. Θα πρέπει λοιπόν στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διατεθούν με τρόπο πιο ευφυή οι υπάρχουσες μορφές χρηματοδότησης. Έχουμε ένα νέο ταμείο στρατηγικών επενδύσεων που παρέχει τεράστιες ευκαιρίες και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε και το κόσμο και τα διαφορετικά ταμεία. Παραδείγματος χάρη 5 Απρίλη έχουμε διοργανώσει μια διάσκεψη για αυτά τα θέματα από την Κομισιόν μαζί με τις τουριστικές οργανώσεις, όλοι είστε προσκεκλημένοι βέβαια και η αγορά των κεφαλαίων μας έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευκολότερη για τις επιχειρήσεις και να χρηματοδοτούνται πιο εύκολα. Δεξιότητες. Τους επόμενους μήνες, το Μάη, θα, θα δημοσιεύσουμε ένα θεματολόγιο δεξιοτήτων. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή εδώ στις υψηλές δεξιότητες που χρειάζονται σε ένα εξειδικευμένο τομέα όπως ο τουρισμός. Επίσης ένας τρόπος με τον οποίο το δημόσιο θα μπορούσε να βοηθήσει είναι η αφαίρεση φραγμών και εμποδίων και η εφαρμογή της στρατηγικής της ενιαίας αγοράς που υιοθετήθηκε μόλις τον Οκτώβρη. Αναφέρθηκα και στη σημασία των μικρομεσαίων για τον τουρισμό ώστε να αντιμετωπίσουμε σωστά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουριστικός τομέας. Επίσης, σας ανέφερα προηγουμένως και τα πλεονεκτήματα τη συνεργατική οικονομία. Πρέπει να γνωρίσουμε ότι κάποιε παρουσιακέ μορφέ επιχειρήσεων φοβούνται ότι αυτέ οι νέε επιχειρήσει θα εκμεταλλευτούν θέματα εργασιακά ή φορολογικά κτλ. Καταρχά λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε και να προσφέρουμε σαφήνεια σε αυτές τις επιχείρησεις. Θα το συζητήσω και αλλού σε άλλες επιτροπέ αυτό το ζήτημα, αλλά να σα πω από τώρα ότι μέσα στο έτος, στις αρχές του Ιούνιου πιθανώς, θα εκδώσουμε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των, της τονής νομοθεσίας. Δεν θέλουμε λοιπόν νέα νομοθεσία, αλλά θέλουμε ξεκάθαρες ή πιο σαφείς κατευθύνσεις για το πώς ακριβώς μπορεί να εφαρμοστεί η υπάρχουσα νομοθεσία σε σχέση με την συνεργατική οικονομία. Αυτό πρέπει να, πρέπει να είναι σαφές σε όλους. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, ε, να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον, να βοηθήσουμε την εφορία και βεβαίω να προστατεύσουμε του καταναλωτές. Σε όλα αυτά δεν μπορούμε να δράσουμε μόνοι μας, χρειαζόμαστε την βοήθεια των χωρών μελών. Πρέπει να δράσουν ώστε να αφαιρεθούν τα περιττά εμπόδια και η γραφειοκρατία και αυτό θα πρέπει να γίνει με ενιαίο τρόπο. Μετά θα πρέπει να βοηθήσουμε τι επιχειρήσει να συνεργαστούν με άλλε δημόσιε αρχέ για την πρόθεση τη Ευρώπη. Συνεργαζόμαστε με την UNESCO, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο για μια κοινή πρόθεση. Στοχεύουμε σε αγορέ τρίτων χωρών, ΗΠΑ, Κίνα, Νότια Αμερική και ενδεχομένω και άλλε ανερχόμενε αγορέ όπω η Ινδία χρησιμοποιούμε θέματα όπως η μόδα, η γαστρονομία, η κληρονομιά. Συνοψίζοντας, νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς σήμερα βέβαια να απεσιοδοξεί για τον τουρισμό. Εγώ διαφωνώ. Θα πρέπει να δράσουμε και το λέω παντού όπου και να βρίσκουμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε, θα πρέπει να δράσουμε από κοινού. Η Κομισιόν θα πρέπει να είναι βέβαια ενεργή στο να προετοιμάσει το περιβάλλον, το κατάλληλο, αλλά οι χώρε μέλη στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο, αλλά και οι τουριστικέ οργανώσει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι όλοι ενεργοί στο να εφαρμοστούν όλα αυτά και να δώσουν την κατάλληλη καθοδήγηση και να προσφέρουν ιδέε. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ενισχυθεί όλο και περισσότερο ο ευρωπαϊκός τουρισμός, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τις θέσεις εργασίας που χρειάζεται πάρα πολύ η πυρός μας και η Κομισιόν είναι δεσμευμένη στο να βοηθήσει τους πάντες για να το πετύχουμε αυτό. Και θα το κάνουμε δημιουργώντας ευκαιρίες όπως έλεγα, αφαιρώντας φραγμούς και συνεργαζόμενοι όλοι μεταξύ μας με όλους τους ε, φορείς του κλάδου αυτού, γιατί πραγματικά αυτό αποτελεί μια ουσιώδη εταιρική σχέση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία και τώρα έχει το λόγο ο πρόεδρος της ειδική ομάδας για τον τουρισμό. Κουρ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για μας ε, που καλωσορίζουμε εδώ την Επίτροπο με αυτή την ευκαιρία και χαιρετίζουμε τα όσα είπατε. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, πρόκειται για μια σημαντική πολιτική απόφαση και είναι πραγματικά ενδεδειγμένη χρονική στιγμή που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης που ήρθατε στη συνάντηση του Task Form. Φως. Είστε πολύ σημαντικό πρόσωπο για μας γιατί δεν έχουμε κανένα άλλο συνομιλητή που μπορεί να μας ε, βοηθήσει ε, και ο οποίος μπορεί πραγματικά να υπερασπιστεί ανά πάσα στιγμή το τουρισμό. Άρα είναι δεδεμένη στιγμή, είναι μια σημαντική καμπή και όπως είπατε κυρία Επίτροπε ε, μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι έχουμε όλα αυτά τα εξαιρετικά δεδομένα που αφορούν το τουρισμό, αλλά είναι το αποτέλεσμα επιτευμάτων του παρελθόντος. Ε, και αν δεν ε, πάρουμε κάποιες αποφάσεις, υποστηρίξουμε τις αποφάσεις με το σωστό τρόπο, φοβούμε, για παράδειγμα σε πέντε χρόνια δυστυχώς, θα καταλήξουμε μη ανταγωνιστική στον τομέα του τουρισμού. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι αυτό που θέσετε στην αρχή. Στο Κοινοβούλιο έχουμε μια επιτροπή, μια ειδική ομάδα και η δική μας ομάδα έχει το καθήκον να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Όχι σαν ένα είδος ε, τυχαίο χόμπι, αλλά είναι πραγματικά το καθήκον μας να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας στο κλάδο τουρισμού και όλους τους εργαζόμενους σε αυτό το κλάδο. Και πάλι λοιπόν, σας καλωσορίζω κυρία Επίτροπε. Ο κύριο Κράμερ στα εισαγωγικά του σχόλια ανέφερε ότι από το 2014, από το 2013 συγγνώμη, είναι αυτή η πρώτη φορά που συναντούμε μια επίτροπο αρμόδια για αυτό το χαρτοφυλάκιο. Είναι σημαντικό λοιπόν για μας. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που ήρθατε εδώ. Είναι σημαντικό θέμα και αυτό μας το καταδεικνύει το γεγονός ότι έχουμε 17 ε, σημαντικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στον κλάδο του τουρισμού, 17 στο σύνολό τους ε, και ε, ίσως πέρσι το φθινόπωρο όταν ο ο οργανισμός τουρισμών, τουρισμού των Εθνών συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του ΠΟΕ, ήταν μια μεγάλη διοργάνωση αλλά πραγματικά είναι μια σημαντική στιγμή για μας. Είναι σημαντικό να συνεργαστούμε και θα ήθελα να σας επισημώνω τρία σημεία. Κύριε Πέτροπε, στην αρχή της ομιλίας σας αναφέρατε κάτι το οποίο ήταν τέλος σημαντικό, το γεγονός ότι δεν έχουμε πολλά νομικά εργαλεία όσον αφορά την υποστήριξη του τουρισμού. Συμφωνώ μαζί σας. Χρειαζόμαστε αυτό το οποίο θα θέλαμε είναι να έχουμε κάποια υποστήριξη, ουσιαστική υποστήριξη για αυτό τον κλάδο. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η φωνή μας ακούεται και εσείς ε, θα είστε η δική μας ε, εκπρόσωπος. Γιατί πραγματικά είστε στο κατάλληλο πρόσωπο. Επίσης χαρίζει το γεγονός ότι αναφέρατε μία έκθεση της ε, συναδέλφης Αβαλνταλμούντα η οποία ε, προετοίμασε αυτή την έκθεση η οποία συζητήθηκε στο Κοινοβούλιο. Σε ευχαριστούμε επίσης και για την δική σας απόκριση ότι πράγματι ο τουρισμός για την Ευρώπη είναι ένας πολύ σημαντικός ε, κλάδος. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πώς εξηγείτε ότι δεν έχουμε ούτε ένα κείμενο της Επιτροπής Juncker που να αναφέρεται στον τουρισμό. Γιατί στο σχέδιο Juncker δεν γίνεται απολύτως καμία μνήα του τουρισμού. Γιατί δίδονται τόσο πολλά χρήματα σε άλλες ε, προτεραιότητες και παραμελείται εντελώς ο τουρισμός. Τι γίνεται για το γεγονό ότι ο τουρισμός πραγματικά παρέχει θαυμάσια ευκαιρίες κατά της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Πώς γίνεται να μην εμφανίσετε πουθενά στα κείμενα της Επιτροπής. Κυρία Επίτροπε, στην ομιλία σας, αυτό το οποίο είπατε είχε σε πραγματικά θαυμάσια στα αυτιά μας. Το χαιρετίζουμε και ελπίζουμε το μήνυμα αυτό να περάσει. Και θέλουμε πραγματικά να είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά ακούγονται από, το, από όλους στην, Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρθηκατε στην, ε, στον εργό ρόλο της Επιτροπής, ε, στο γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ενεργητικότητα και δυναμισμός. Επίσης από τις ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις. Υπάρχουν δύο θέματα που θα ήθελα να ευθύνω σας κυρία Επίτροπε. Καταρχήν, βλέπετε καμία ευκαιρία για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τουρισμού Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση από το Συμβούλιο. Δεύτερο ερώτημα. Θα ήθελα να μας πείτε για τη διαδικασία αυτή ε, του μεταξύ Ηνωμένων Εθνών και ΠΟΕ. Ο κύριος, η κυρία Τσαπατέλ ε, αναφέρθηκε σε αυτή τη συνεργασία στο Intergroup. Το 2018 θα είναι το έτος του Ευρωπαϊκού Τουρισμού και προωθήθηκε η ιδέα αυτή. Πώς, σε ποιο βαθμό έχουμε προχωρήσει, πώς μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα τη συνεργασία μας. Κύριε Επίτροπε και πάλι σε ευχαριστούμε για την ανάλυση σας, γιατί στη βάση όλων αυτών μπορούμε πραγματικά να συνεργαστούμε πολύ καλά στο μέλλον και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι από τις διάφορες πολιτικές ομάδες θα, με, θα μας υποστηρίξουν. Η κυρία E, e, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι πολύ που είναι σήμερα εδώ η Επίτροπος. Συμφωνώ με τους συναδελφούς. Ο τουρισμός είναι όντως ένας πολύ σημαντικός κλάδος της οικονομίας. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό και γνωρίζουμε και την ανάγκη που υπάρχει να αυξηθεί ο τουρισμός προς την Ευρώπη. Αλλά πρέπει να δούμε και τα γεγονότα του Παρισιού και πώς αυτά έχουν επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό. Γιατί πολλοί θα επιλέξουν κάποιο διαφορετικό μέρος για να πάνε να κάνουν τις διακοπές τους. Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη και την οικονομική διάσταση. Η... Τα ταξιδιωτικά γραφεία που ε, δραστηριοποιούνται στο Παρίσι, σε άλλες ε, πόλεις όπου υπάρχουν ε, τέτοιου είδους συμβάντα, όπως οι δημοκρατικές επιθέσεις, επηρεάζονται αρνητικά. Ένας τρόπος για να αποφύγει κανείς τέτοιου mm. είδους καταστάσεις και να εξασφαλίσει ότι οι τουρίστες ας πούμε από την Ασία ή από την Αμερική θα έρθουν προς την Ευρώπη είναι να προωθήσουμε τον κλάδο αυτό. Δυστυχώς στο σχέδιο Juncker δεν βλέπουμε κάποια οικονομικά μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ίσως για τον, από τον κλάδο αυτό. Τον πολύ σημαντικό κλάδο για την οικονομία και έναν κλάδο ο οποίος ε, επηρεάζει θετικά την ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η Ζαμπέλα Ντεμόντε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω και εγώ και να καλωσορίσω την Επίτροπο. Είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά που είναι μαζί μας σήμερα και ήδη είπε ότι θα είναι διαθέσιμη για συζητήσεις και αυτό πραγματικά δείχνει την αφοσίωση που δείχνει στον κλάδο του τουρισμού. Ε, υποστηρίζω πλήρως να πω το ότι ο τουρισμός θα πρέπει να θεωρηθεί βιομηχανία. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε ουσιαστικά δίνουμε μια δικαιολογία στον εαυτό μας για να μην δώσει την δέουσα προσοχή σε έναν κλάδο ο οποίος συμβάλλει πάρα πολύ σημαντικά στο καθάριστο εθνικό προϊόν. Ε, νομίζω επίσης ότι πρέπει να υπάρξει και ένα σχέδιο δράσης. πρέπει να δούμε τον μελλοντικό προγραμματισμό. Και επίσης να θέσω ένα ερώτημα. Πώς θα θέλατε να προωθηθεί η έκθεση πρωτοβουλίας, ε, για ποιους ε, κλάδους, με ποιους στόχους ε, θεωρείτε ότι μπορούν να αποτελέσουν κλειδιά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς βεβαίως έχουμε το δικό μας ρόλο να παίξουμε, αλλά εσείς από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρείτε ότι θα μπορούσε ίσως ας πούμε, ο τουρισμός να αποτελέσει κομμάτι ή αντικείμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης. Ε, δεν είναι απόλυτα σαφές που εντάσσεται ο τουρισμός ε, στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως να πρέπει να γίνει πιο ορατός και ίσως ε, θα πρέπει όσα αφορούν στον τουρισμό, δηλαδή πληροφορίες, να είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες. Οι πληροφορίες και το εγχειρίδιο για τα κονδύλια τα οποία αποδίδονται στον ε, κλάδο του τουρισμού. Θα πρέπει να υπάρχει αποδοτικότητα, ε, επάρκεια ό,τι αφορά τους πόρους. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφόρηση σχετικά. Και επίσης, στο παρελθόν έχουμε συζητήσει για τον ε, θαλάσσιο και τον παράκτιο τουρισμό. Ίσως και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας ειδικός κλάδος του τουρισμού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λουτόφσκι έχει το λόγο. Να καλωσορίσω και εγώ την Επίτροπο στην Επιτροπή μας. Τρία ερωτήματα έχω να θέσω. Ο ψυχολογικός τουρισμός, ε, τα ΣΠΑ επίσης. Το θέμα αυτό δεν έχει τύχει της απαραίτητης προσοχής. Δεν έχει μελετηθεί εις βάθος. Επίσης, βλέπετε μήπως ε, κάποια δυνατότητα ανάπτυξης του τουρισμού σε λιγότερο ελκυστικές περιοχές, γιατί τα σπα, όπου και να είναι, είναι ελκυστικά από μόνα τους. Επίσης, ένα ψήφισμα για την ε, δημιουργία του Ευρωπαϊκού Εμβλήματος Ποιότητας. Για περιοχές που είναι φιλικές προς τις οικογένειες. Αυτό βοηθάει καθόλου προς την κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε, αρκεί ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης, αυτά που, σε σχέση με αυτό που είπε ο συνάδελφος, έχετε κάποια πληροφόρηση για την επιρροή για τον αντίκτυπο της προσφυγικής κρίσης στο, στην βιομηχανία του τουρισμού στην Ευρώπη, ειδικά σε ό,τι αφορά τον κύκλο σε χώρους όπου υπάρχουν ε, πρόσφυγες. Ελέγχετε την κατάσταση, έχετε κάποιες εναλλακτικέ λύσεις, ε, πιστεύω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στις, στους προορισμούς που επιλέγονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η επό... επόμενα είναι η κυρία Μπαραντίκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε για την παρουσίαση των... του προγράμματός σας. Και θα ήθελα να σας αναφέρω δύο θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι αναγκαίο ε, να δούμε στον τομέα, στον κλάδο του τουρισμού στην Ευρώπη και να προετοιμαστούμε για αυτή την ανάπτυξη η οποία έχει προβλεφθεί σε αυτές τις ε, μελέτες αντικτύπου περισσότεροι από 8 εκατομμύρια τουρίστες ε, τα επόμενα χρόνια και νομίζω θα πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Η ψηφιοποίηση είναι σημαντική για, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και νέων βιομηχανιών. Και θα ήθελα να σας πω ότι στη χώρα των Βάσκων για το 2015 ζούσαμε αριθμούς ε, ρεκόρ πάνω από 3 εκατομμύρια τουρίστες, κάτι το οποίο δεν ήταν συνηθισμένο στη δική μας ε, περιοχή. Το 70% των τουριστών που μας επισκέπτονται το κάνουν μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας που το κάναμε για να προβάλλουμε τον τουρισμό μας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Εσείς αναφερθήκατε στις ευκαιρίες που έχει ο τουρισμός για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε εάν στο επίπεδο της Επιτροπής έχετε προβλέψει να καταρτήσετε, να κάνετε κάποια δουλειά ε, σε εγκάρσια, γιατί ε, ο τουρισμός συνεπάγεται την ανάγκη εκτέλεσης των ευρωπαϊκών ε, προγραμμάτων, προγραμμάτων προτεραιότητας, ούτως ώστε να βελτιώσουμε και τα προγράμματα απασχόλησης για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία που υπάρχει σε ορισμένες νέες χώρες. Μέσω αυτής της νέας πιθανότητας που αντιπροσωπεύει ο τουρισμός. Και το θέμα των πανεπιστημίων είναι επίσης ε, καθοριστικό για να δοθεί μια πιο σφαιρική, ε, υπάρξει μια πιο σφαιρική προσέγγιση θα πρέπει να υπάρχει για τους ανθρώπους αυτούς μια πανεπιστημιακή κατάρτιση με γλώσσες, ε, εκπαίδευση γλωσσών κλπ. Και επίσης αναφερθήκατε στην συνεργατική οικονομία σαν ε, μια καινοτόμα εξέλιξη. Θα ήθελα να μας πείτε το εξή. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάθε χώρα έχει τη δική της ε, προσέγγιση. Ε, όσον αφορά αυτό το εγκάρσιο μοντέλο, όπου πιστεύω θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο... να υπάρχουν μεγαλύτερα αποτελέσματα. Γιατί υπάρχουν και άλλες ε, πλατφόρμες για την εξέλιξη στον κλάδο του τουρισμού. Πιστεύετε ότι θα μπορεί να υπάρξει εδώ, να γίνει ένα ακόμα βήμα. Ευχαριστώ κυρία Τζιλ um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, συγγνώμη που έχασα την εισαγωγή και ήρθα αργά. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, χαιρετίζω αυτά που είπατε σήμερα ιδιαίτερα την έμφαση στην εκμάθηση, στις δεξιότητες, στους νέους που για αυτούς που εκπροσωπώ εγώ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς αναπτύξαμε ένα επιτυχές πρόγραμμα υπαίθρινων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στο βορρά της χώρας, κάτι το οποίο προσέλκυσε πολλούς νέους και είχαμε έτσι ένα νέο κοινό και μια νέα πλατεία από όλο τον κόσμο. Έχουμε και θέματα βέβαια μεταφορών και προβλήματα, αλλά νομίζω ότι σωστά δίνεται συγκεκριμένη έτσι στόχευση. Κατευθυντικές γραμμές που αναφέρατε, δηλαδή η σύνδεση τουρισμού και του πολιτισμού, είναι ευπρόσδεκτα. Τώρα τα πρωτόκολλα τουρισμού και μεταφορών είναι πολύ σημαντικά μια σύμβαση των Άλπαιων για την προώθηση του τουρισμού στις Άλπεις. Να σας ρωτήσω όμως εγώ κάτι σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από τα Ταμεία Συνοχής και τα Περιφερειακά Ταμεία, ας πούμε τουριστικά προγράμματα, γιατί σε πολλές περιοχές όπως τη δική μου θα πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομία και οι περιοχές που λαμβάνουν κονδύλια από περιφερειακά και ταμεία συνοχής. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη όλα αυτά. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε αιτήσει ανασκοπήσεις όλων αυτών των προγραμμάτων στον με την αποτελεσματικότητά τους. Ευχαριστώ. Κυρία συγγνώμη που καθυστέρησα κι εγώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε για να μιλήσουμε για ένα τομέα ο οποίος μας ενδιαφέρει πολύ. Λυπάμαι που απουσιάζουν πολλοί συνάδελφοι κιόλα. Εγώ κατάγομαι από το νότο της Ιταλίας, δηλαδή μια από τις περιοχές που έχουν λιγότερη, χαμηλότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τον τουρισμό. Ίσως λόγω και μια σύγχυσης που υπάρχει, επειδή δεν υπάρχουν πολλά κονδύλια άμεση χρηματοδότηση που αφορούν τον τουρισμό. Κάποιο πρέπει να ψάξει λίγο, να τα αναζητήσει τα κονδύλια αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω γιατί δεν υπάρχει πάνω στο θέμα αυτό σαφήνεια εκ μέρου τη Κομισιόν. Υπάρχει μεγάλη ησυχή, στο ξαναλέω. Θα πρέπει να υπάρχει ένα προνομιακό κανάλι χρηματοδότηση. Γιατί όλα αυτά να εντάσσονται ας πούμε, στα προγράμματα που αφορούν τι μικρομεσαίε, θα μπορούσε ενδεχομένω να δυσκολέψει ένα τομέα που παρουσιάζει πολλέ ιδιαιτερότητε. επειδή πολλοί τομεί είναι εποχιακοί δεν εργάζονται όλο το χρόνο οπότε σε σχέση με άλλου τομεί με μικρομεσαίε που εργάζονται 12 ε, μήνε, τότε ίσω να έχουμε κάποια ανισότητα ρωτάω λοιπόν από τη στιγμή που υπάρχουν περιοχέ τη Ευρώπη που δεν έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια. Έχετε στρατηγική να βοηθήσετε ώστε αυτό το κενό να καλυφθεί. Γιατί νομίζω δεν βοηθάει κανένα το να διαθέτουμε κονδύλια τα οποία τελικά βοηθούν τους πιο έξυπνους που εκμεταλλεύονται πόρους εις βάρος άλλων περιοχών που έχουν μεγάλο δυναμικό αλλά που δεν καταφέρνουν να δημιουργήσουν πλούτο από αυτό που διαθέτουν έχοντας πάντοτε έτσι κατά νου το νότο της Ιταλίας. Οπότε ποιες στρατηγικές διαθέτει η Κομισιόν για να ξεπεραστεί αυτή η τεράστια δυσκολία που υπάρχει και που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι στον κλάδο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Okay, good. Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Δεν είμαι απεσιόδοξη. Εγώ είμαι αισιόδοξη για το μέλλον του τουρισμού. Εγώ είμαι από την Ιρλανδία. Τα πράγματα είναι πολύ θετικά εκεί και νομίζω ότι αυτό έχει συμβάλει και πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις της ενεργείας. Έχουμε τη μεγάλη αύξηση στον τομέα αυτό, των θέσεων εργασία που υπάρχουν. Για τη συνεργατική οικονομία τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε ένα σημείο που θα έχουμε κάποιες διευκρινήσεις και, θέσεις, και κάποιες κατευθυντήρες γραμμές, γιατί ο χρόνος περνάει, η τεχνολογία προχωράει και βλέπουμε τις προκλήσεις και την ε, έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει ε, προς τους διάφορου παρόχους υπηρεσιών και νομίζω ότι πρέπει αυτό το θέμα να το λύσουμε, να μην αφήσουμε τα πράγματα να λιμνάζουν έτσι. Υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει τεχνολογία, οι καταναλωτές την χρησιμοποιούν και όλο και περισσότεροι καταναλωτές έχουν ένα iPad ή ένα iPhone και κάνουν μόνοι τους τις, ε, ε, οργανώνουν μόνοι τους τις ε, διακοπές τους και τα ταξίδια τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα έχουμε ένα ξεκάθαρο τοπίο έτσι ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. ορίζω λοιπόν τα σχολεία σας σχετικά. Να ρωτήσω επίσης για το σήμα ποιότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού που αναφέρεται στην έκθεση, στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Τι έχει γίνει με αυτό η εφαρμογή επίσης του, της ανακοίνωσης του 2010 για τον τουρισμό. Υπάρχει μια μελέτη σχετικά, ε, σας βοήθησε να χαρτογραφήσετε λίγο τις αποφάσεις για το μέλλον και επίσης οι συγκεκριμένες ε, ε, ε, προκλήσεις για τον παράκτιο τουρισμό. Αυτή είναι όντως σημαντική πρόκληση σε ό,τι αφορά και τη διασύνδεση των νησιών και τις υπερπεριφερειακές περιοχές. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να προχωρήσει. Είναι νομίζω ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά της, ε, που αντιμετωπίζουν τέτοιες περιοχές ε, σε ό,τι αφορά τη διασύνδεσή τους. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Επίτροπε. Θεωρώ ότι η συνάντησή μας εδώ αυτή είναι ευτυχής είναι κάτι που μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε με καλό τρόπο τη συζήτηση για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Στη θητεία μας αυτή θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δει τη γέννηση μιας ε, σημαντικής κίνησης, ενός ρεύματος με τη δημιουργία μιας ε, ομάδας ενδιάμεσης, ένα intergroup, μιας task force για, το, για την κληρονομιά κτλ. Αυτές οι δύο δομές που έχουμε δημιουργήσει χρειάζονται περισσότερη προσοχή, χρειάζονται περισσότερη βοήθεια πολιτική για τον τομέα αυτό που όπως ξέρουμε όλοι διαδραματίζει βασικό ρόλο για την ευρωπαϊκή οικονομία που όχι μόνο θα πρέπει να παραμεληθεί αλλά να παροτρινθεί και να ενισχυθεί. Θέλουμε, Επίτροπε, σχέσεις πιο στενές για να συζητάμε τα προβλήματα του τουρισμού. Θέλω λοιπόν να επωφεληθώ αυτή της ευκαιρία της παρουσίας σας εδώ, σήμερα στην Επιτροπή μας. Να επωφεληθώ λοιπόν της ευκαιρία αυτή που έχουμε σήμερα για να πω ότι εδώ έχουμε και συναδέλφους που είναι βέβαια μέλη σε άλλες επιτροπές εκτός από τη δική μας. Και οι επίτροποι, οι συγγνώμη συνάλφοι αυτοί γνωρίζουν ότι υπάρχουν και οργανώσει του τουρισμού οι οποίοι μέχρι τώρα μας συνόδευσαν, μας βοήθησαν από τότε που ξεκινήσαμε τη θητεία μας στο Κοινοβούλιο, με τους οποίους συνεργαστήκαμε με τους οποίους καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια καλή σχέση ώστε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Καταρχάς, χρειαζόμαστε περισσότερη χρηματοδότηση με καλύτερο συντονισμό για τις μικρομεσαίες του τουρισμού. Όπως ξέρετε κι εσείς, αλλά και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο, ο ο υπολογισμός το 16 για τον τουρισμό έχει μειωθεί και αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια επειδή εμεί θα επιθυμούσαμε να υπάρχουν συγκεκριμένε προτάσει από την Κομισιόν μέσω του προσώπου σα ή μέσω του κυρίου Γιούνκερ ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού με το σχέδιο Juncker. Εσείς αναφερθήκατε στι δυνατότητε που υπάρχουν, όμω, αυτέ οι δυνατότητε θα πρέπει να γίνουν πιο απτέ, πιο συγκεκριμένε στο ταχύτερο δυνατό, ώστε να υπάρχουν σαφές, λύσει και ένα σύστημα με το οποίο θα διασυνδέσουμε τι μικρομεσαίες του τουρισμού με το σχέδιο του Juncker. Κάτι άλλο, η γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία θα πρέπει να περιοριστεί όσο γίνεται, ώστε να αναπτύξουμε και τον τουρισμό στι ευρωπαϊκέ περιφέρειε. Ξέρετε ότι Θέλουμε να έχουμε μια νέα στρατηγική για τον τουρισμό και μιλώντας με εσά όμως κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι θέμα προτεραιότητας για την Κομισιόν προς το παρόν τουλάχιστον. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το ταχύτερο δυνατόν να διαθέτουμε ένα σχέδιο δράσης με αξιολογήσεις, με αναλύσεις και με κατευθυντήριε γραμμέ. Αν κάνουμε αυτή την αξιολόγηση, τότε θα καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να βελτιωθούν στον ευρωπαϊκό τουρισμό, ώστε να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο παρέμβαση εκεί ακριβώ που μα επιτρέπουν τα υπάρχοντα εργαλεία. Τώρα βέβαια δεν θέλω να ξεχάσω και του εταίρου μα από τον τομέα του τουρισμού, οργανώσεις, ιδιωτικέ επιχειρήσει κτλ. που μαζί έχουμε συντάξει αυτό το μανιφέστο για την απασχόληση και τον τουρισμό όπου περιγράφονται ακριβώ τα υπέρ κατά αυτού του τομέα. Είναι λοιπόν σημαντικό να ακούσουμε του φορεί και είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε μια καλά συντονισμένη δομή για το μέλλον του τουρισμού που θα βασίζεται και θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα του ιδιωτικού τομέα. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε και μια εταιρική σχέση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιωτικό τομέα του τουρισμού και νομίζω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να αποτελέσει ένα μόνιμο εταίρο στην δομή αυτή. Επίσης, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το δεχόμενο ευρωπαϊκής χρονιάς τουρισμού για το 2018. Α, θα γνωρίζετε ότι το 2017 είναι το έτος βιώσιμης ανάπτυξης τουρισμού, όπως ανακηρύχθηκε από τον ΟΙΕ. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε κάτι αντίστοιχο από το Κοινοβούλιο και θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό έτος τουρισμού. Ήδη από πέρσι σας προβάλαμε το αίτημα αυτό και ζητάμε να υποβληθεί επίσημα προς το Συμβούλιο αυτό το αίτημα ώστε να ανακηρυχθεί το 2018 επίσημο έτος τουρισμού και ανάπτυξης. μάλιστα και ο ΙΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει και να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία για την στήριξη δηλαδή, του ευρωπαϊκού τουρισμού. Τώρα, όσον αφορά την προώθηση ε, λιγότερο γνωστών προορισμών, τουριστικών προορισμών στην Ευρώπη, εμείς θεωρούμε, εμείς θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε κάποια πράγματα σε επίπεδο marketing υπέρ αυτών των λιγότερο γνωστών περιοχών διευκολύνοντας ή προβάλλοντας τις μεταφορές, την σύνδεση με αυτά τα μέρη. Οπότε ε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ενδεχομένω και ένα σήμα αριστείας ευρωπαϊκού τουρισμού που θα βοηθήσει ακριβώς τις λιγότερο γνωστές περιοχές, τους λιγότερο γνωστούς ε, προορισμούς να αναδειχτούν, όπως στη Ρουμανία αλλά και σε άλλες χώρες. Το έχουν αναφέρει αυτό και άλλοι υπουργοί τουρισμού των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης ε, περιοχών, γεωγραφικών περιοχών με πολύ καλά τοπία, με αναπτυγμένο ε, με αναπτυγμένη πολιτιστική διάσταση κλπ. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν το λόγο είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή ιδιαίτερη σε αυτά τα ζητήματα. Εμείς πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε και στο μέλλον μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τον τουρισμό. Αυτή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τον τουρισμό πιστεύω θα μπορούσε να στηρίξει και μια Ευρωπαϊκή Ακαδημία για την ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων στον τουρισμό, γιατί στον τομέα του τουρισμού χρειαζόμαστε ιδιαίτερες δεξιότητες, ακριβώς για να ενισχύσουμε και να αυξήσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει ο τουρισμός και να βοηθήσουμε την διεθνή του ανταγωνιστικότητα. γιατί είναι αλήθεια ότι η διεθνής αγορά του τουρισμού είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Ζητώ συγγνώμη αν μακριόρισα, λέει μιλήτρια. Είναι πάρα πολλά τα αιτήματα που έχουμε. και αυτό μπορούσε να κάνει το Κοινοβούλιο για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού. Όχι μόνο λόγω του πάθους που έχουμε για αυτό τον κλάδο, αλλά λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας ο τουρισμός, αλλά και για την ανάπτυξη βεβαίω των οικονομιών των μεμονωμένων κρατών μελών. Σας ευχαριστώ πάντως που ήρθατε σήμερα εδώ και ελπίζω να εκφράσω το σύνολο των αδέλφων λέγοντας ότι ελπίζω ότι θα μπορούμε να βρούμε σε εσά και στον κύριο Γιούνκερ ένα αξιόπιστο εταίρο για την ανάπτυξη του τουρισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έβαλα και πάλι το όνομά μου στον κατάλογο. Βεβαίω, ο, ο τουρισμός Also, ich Έγραψε το όνομά μου στον κατάλογο. Ο τουρισμό βεβαίω έχει μια οικονομική πτυχή, την οποία φυσικά αναφέρατε και βεβαίω ξέρουμε από την εμπειρία μα ότι ο τουρισμό μπορεί να καταστρέψει τον τουρισμό. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μιλήσω για τον ποδηλατικό τουρισμό που αυξάνεται 20% κάθε δύο χρόνια. Ε, οι περισσότεροι ήταν φοιτητέ και χαμηλών εισοδημάτων άνθρωποι. Ξέρουμε ότι τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ε, ξέρουμε πολλού που έχουν τη Mercedes στον καράζ του και παίρνουν το ποδήλατο και κάνουν ταξίδια. Ε, και μάλιστα ένας ε, ταξιδιώτης ε, ξοδεύει 35 ευρώ τη μέρα όταν κάνει διακοπές με το ποδήλατό του, ενώ ένα που πάει με το αυτοκίνητό του μόλις 10 ευρώ. 44 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανώνται κάθε χρόνο από το, αυτού του είδους του τουρισμού όπως και από τις κρουαζιέρες. Το να πάρουμε 10-15 εκατομμύρια από τους ποδηλάτες για να τους προστατεύσουμε και να τους προωθήσουμε είναι δύσκολο. το να, να λάβουμε πολύ περισσότερα χρήματα από άλλου είδους τουρισμού είναι πολύ, είδη τουρισμού είναι πολύ εύκολο. Ε, πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε και αυτόν τον κλάδο τουρισμού που, είναι, που έχει πολύ μεγάλο οικονομικό ε, αντίκτυπο. Υπάρχουν πολύ περισσότερες ε, βιομηχανίες κατασκευής ποδηλάτων στην Ευρώπη, αλλά δεν παίζουν τον ρόλο που του αναλογεί. Και επίσης έχουμε το πρόβλημα ο τουρισμός να εξαρτάται από την εποχή. Ε, πήγαμε στη Φιλανδία με την Επιτροπή. Βεβαίω, το χειμώνα, ο τουρισμός στη Φιλανδία είναι ωραίο πράγμα. Αλλά μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει κάποια μονοπάτια το καλοκαίρι ως ποδηλατόδρομους. Ε, δεν το ξέραμε, το είδαμε και το καταλάβαμε. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ θετική, έχει πολύ θετικό αντίκτυπο. Το κάνει και η Αυστρία και η Ελβετία επίσης. Είναι σημαντικός λοιπόν ο, ο τουρισμός. Δεν χρειάζεται πολλά ε, χρήματα για την υποδομή, αλλά τα ωφέλη είναι πάρα πολλά ίσως καλό θα ήταν να υπάρχει και μια πιστοποίηση για βιώσιμο τουρισμό, ε, γιατί ξέρουμε ότι ε, καταγράφεται κάπου ότι είναι βιώσιμο ο τουρισμό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Ίσως λοιπόν να χρειάζεται μια διαδικασία και γι' αυτό βλέπετε μια δυνατότητα να υπάρχει μια καλύτερη υποστήριξη. Και να δώσω τώρα το λόγο στον Πασκάλ. Έχω σημειώσει τους πάντες, μη στεναχωριέστε. Ε, είσαστε στον κατάλογο, οπότε ήρθε η σειρά σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Συνήθως μιλώ τελευταίος. Πρόεδρε και Επίτροπε, είμαι εδώ από τις 9 το πρωί, κάναμε δύο διαλύματα Μετά οι αλκυστήρες μάλλον ευφύ λένε ότι είναι αλλά δεν είναι και τόσο, οπότε φτάσαμε αργά. Καστήρισαμε. Έχασα λοιπόν την εισαγωγή σας, αλλά φαντάζομαι ότι θα ήταν ενδιαφέρουσα. Κυρία Επίτροπε, εδώ στην Επιτροπή μας είμαι 11 χρόνια και μιλάω συνέχεια για το θέμα του τουρισμού. Είμαστε Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού δεν είναι ίσον σημασία ο τουρισμός. Στην χώρα μου την Ισπανία είναι η καλύτερη επιμηχανία, η μεγαλύτερη πηγή πλούτου και δημιουργίας απασχόλησης. Δημιουργεί πολιτισμό, προβολή, κοινωνικών θεμάτων, έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία. Στο 125 άρθρο λέει η συνθήκη ότι δεν γίνεται να έχουμε εναρμόνιση εδώ σε αυτό το θέμα. Και αυτό με παραξενεύει γιατί η Κομισιόν βασίζεται σε αυτό ακριβώς για να μην νομοθετήσει επαρκώς. Θα ρωτήσω λοιπόν εγώ αυτό, Επίτροπε. Πώς θα μπορέσουμε να συνεπάρξουμε με αυτή την απαγορεύση της αναρμόνισης και ταυτόχρονα να νομοθετήσουμε Τη στιγμή που υπήρχε μεγάλη αντίρρηση για το σχέδιο Γιούνκερ, όχι για τον κύριο Γιούνκερ, αλλά για το σχέδιό του. Πρέπει λοιπόν να αφιστήσουμε την προσοχή σε αυτό το θέμα. Γιατί δεν αφορά μόνο την Ισπανία αυτό. Αν δεν είχαμε τουρισμό, δεν δηλαδή θα ήμασταν πιο φτωχοί. Έχουμε τι αναπτυσσόμενε χώρε που ανταγωνίζονται την Ένωση. Σε όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε λοιπόν ένα νέο φαινόμενο το οποίο έχει σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό χαρακτήρα. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν αυτά που υπόθηκαν. Πολλά από αυτά πολύ σωστά. Ρωτά λοιπόν το εξή. Κατά πόσο θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε αυτή την απαγόρευση για την εναρμόνιση, ώστε να κάνουμε κάποια από τα πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Τέλος, η συνεργατική οικονομία. Επίτροπε. Δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά η συνεργατική δεν μπορεί να αποτελέσει και αθέμητο ανταγωνισμό. Επ' αυτού θα πρέπει να νομοθετήσουμε. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και έλλειψη νόμου, αλλά και παρανομία. Σε σχέση δηλαδή με αυτούς που πληρώνουν φόρους και είναι νόμιμοι στο θέμα του τουρισμού. Έρχονται λοιπόν κάποιοι που σπρώχνουν κιόλα και βγαίνουν μπροστά με τρόπους αθέμητους. Αυτό θα πρέπει να το ρυθμίσουμε. Θα πρέπει να μην ναι. υπάρχει αθέμητο στοιχείο στη συνεργατική οικονομία. Θα πρέπει λοιπόν να μην υπάρχουν φαινόμενα που δεν ρυθμίζονται και που βλάπτουν αυτούς που είναι νόμιμοι και πληρώνουν φόρους. Η συνεργατική οικονομία λοιπόν θα πρέπει να ρυθμιστεί. Είτε έχουμε να κάνουμε με την διαμονή, είτε με τις μεταφορές. Και τώρα ακριβώς βλέπουμε αυτά τα κενά, τα νομοθετικά, να νομοθετούν, να θέτουν στους νομοθετικούς κανόνες και υπάρχει ένα πραγματικό χάος. Χρειαζόμαστε λοιπόν νομιμότητα. Χρειάζεται να καλύψουμε αυτό το κενό και να νομοθετήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Γιατί αυτό έχει ανακύψει ως έντονο φαινόμενο σε όλους τους τοριστικούς κλάδους των χωρών μας. Χαιρετήσω επίση και την στάση σας να λάβετε πολύ σοβαρά αυτό που είναι εκ πρώτης όψεως ίσον σημασίας αλλά είναι πολύ σημαντικό για τον τουρισμό. Σε πολλές χώρες λοιπόν αναπτυσσόμενες ο τουρισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή κοινωνικού και οικονομικού και πνευματικού πλούτου. Στηρίζουμε λοιπόν τις αποφάσεις που θα λάβετε για να μπει ο τουρισμός ακριβώς στη θέση που του αξίζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Serdecznie witam panią komisarz. Chciałbym króciutko Ευχαριστώ. Να καλωσορίσω και εγώ την Επίτροπο. Ε, θέλω δύο πράγματα να πω. Η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στην, ε, στον κλάδο του τουρισμού. συζητούμε πώς εφαρμόζεται η ε, Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ε, Ατόμων με Αναπηρία. Χτες μάλιστα συζητήσαμε σχετικά και ελπίζω ότι θα υπάρξει ένα ενδιαφέρον έγγραφο σχετικά με τα βήματα που πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία, οι Ευρωπαίοι με αναπηρία, να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα που έχουν στην κινητικότητα και να επωφεληθούν από τον τουρισμό και τα όσα προσφέρονται στον κλάδο αυτό. Αυτό το κείμενο που είναι η σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αναφέρει ότι ο τουρισμός ε, πρέπει να είναι ε, προσβάσιμος στα άτομα αυτά και αυτό έχει να κάνει με την προσφορά που υπάρχει. Γιατί πολλές φορές ε, οι προσφορές που γίνονται, γίνονται εκτός της σεζόν, που σημαίνει ότι μεγαλώνει έτσι, επιμικίνεται η σεζόν και αυτό βοηθάει και στην δημιουργία θέσεων εργασία και άρα ενισχύεται αυτό ο κλάδο τη ευρωπαϊκή οικονομία. Άλλο ένα θέμα που θέλω επίση, Πρόεδρε, να θίξω ε, για τη βελτίωση του, ε, του προσφερόμενου τουρισμού στην Ευρώπη. Με βάση τις διάφορες προσφορές που γίνονται, κάποιες ε, εγκαταστάσεις ήταν ε, σημαντικές κάποτε για την ε, βαριά ας πούμε, βιομηχανία, αλλά τώρα ε, μπορούν να τις επισκεφτούν κάποιοι τουρίστες οι οποίοι να ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους τουρισμό. Ίσως λοιπόν μια τέτοια ενίσχυση από την Κομισιόν τέτοιων πρωτοβουλειών να ήταν καλή για να ενισχυθεί και η εσωτερική προσφορά ε, εντός δηλαδή των κρατών μελών. Γιατί κάποιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται και για πράγματα πέραν των, ε, της ωραίας θάλασσας και της ωραίας παραλίας. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα στις 27 Απριλίου να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, τότε που θα οργανώσουμε ένα σεμινάριο για τη βιομηχανική κληρονομιά και τον βιομηχανικό τουρισμό. Και ελπίζω βεβαίω να μπορέσετε να παραβρεθείτε και εσεί στο σεμινάριο αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ρόζα Στάρα Στεραγκούτη, επόμενη. Sí, muchas gracias. Ευχαριστώ. την Επίτροπο για την παρουσίαση που έκανε σχέση με τον τουρισμό που πράγματι είναι μία από τις βασικότερες πηγές πλούτου, ιδιαίτερος στην ε, Ισπανία. Εγώ προέρχομαι από τις Βαλαρίδες νήσους που πραγματικά ο, ο τουρισμός είναι η βασική πηγή πλουτισμού, πλούτου και που μας βοήθησε να ξεφύγουμε από την κρίση. Η τοποθέτησή μου αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Όσον αφορά το τουρισμό, το 2016 ε, ε, ε διατυπώθηκε νέα μας στρατηγική. Ε, ο τουρισμός είναι μια εθνική αρμοδιότητα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίται ε, και σε περιφερειακό επίπεδο. Τι δρα... μελλοντικές δράσεις ε, προβλέπονται για την πρόθεση του τουρισμού τους ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Είναι αλήθεια ότι η Επίτροπος αναφέρθηκε στις δυσκολίες ε, εναρμόνισης, ε, διότι δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Ε, η Επιτροπή επέμεινε σε θέματα, σε να σε θέματα ασφαλείας αλλά πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει μια ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, ούτως ώστε να υπάρξουν, να διατυπωθούν κάποιες ε, προδιαγραφές ποιότητας και να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σήμα τουριστικής ε, ποιότητας. Στις ε, Βαλερίδας νήσους πρόκειται για την, μια παράκτια τουριστική στρατηγική, μια τουριστική στρατηγική για τις παράκτιες περιοχές και αυτή τη στιγμή εκπώνεται μια μελέτη για τις προκλήσεις ε, της ε, βιώσιμης εξέλιξης και θα παρακολουθήσουμε εκ του σύναγκης τα προβλήματα των νήσων αυτών. Εσείς από τη δική σας πλευρά τι πληροφορίες μπορείτε να μας δώσετε. Τα περισσότερα νησιά της Μεσογείου βασίζονται πράγματι στον τουρισμό. Και ο τουρισμός συνδέεται στα νησιά πολύ περισσότερο με την ε, διασυνδεσιμότητα των γεγονότων. Έχει, ε, πρόκειται για μια καθαρή ενεργειακή μορφή και συμβάλλει θετικά στη Ε, τα περισσότερα από αυτά τα νησιά έχουν ένα τουρισμό ε, εποχιακό και νομίζω ότι χρειάζεται μια διαφοροποίηση εδώ, ε, τουρισμό που ασχολείται με την πολιτιστική κληρονομιά, ε, τουρισμό των επιχειρηματιών, εμπορικό τουρισμό κλπ. Και ε, ένα άλλο θέμα αφορά τις καινοτομίες που είναι αναγκαίες ούτως να υπάρξει αύξηση της ανταγωνιστικότητας και να υπάρξουν νέες εφαρμογές, καινοτόμες εφαρμογές. Πού βρισκόμαστε εδώ όσον αφορά το ζήτημα της καινοτομίας. Και ένα τελευταίο θέμα, η προσβασιμότητα. Ο τουρισμός θα πρέπει να είναι ε, προσβάσιμος. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους ηλικιωμένου και στα άτομα με αναπηρία. Ε, Βεβαίω η ομάδα αυτή είναι σημαντική γιατί πρόκειται για 80 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη που εντάσσονται εδώ και όταν κανείς ε, θέλει να αγοράσει ένα τουριστικό πακέτο, το, ε, το άτομο με... Ε, που είναι περισσότερη κινητικότητα πρέπει να γνωρίζει το επίπεδο της προσβασιμότητας. Για να μην υπάρχουν προσδοκίες που τελικά διαψεύδονται όσον αφορά την προσβασιμότητα. Εγώ δεν αναφέρομαι στην προσβασιμότητα των ε, ξενοδοχείων μόνο, αλλά για παράδειγμα των ε, δυνατοτήτων αθλητισμού. Άρα λοιπόν η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντική εδώ. Και τέλος, όλο το, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ το οποίο θα οργανωθεί το 2017. Τι έχουμε να περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομο και να ολοκληρώσω αυτό τον ε, γύρο παρεμβάσεων. Κυρία Επίτροπη, ακούσατε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν πολλές ε, προτάσεις στο τραπέζι, πολλές ιδέες, πολλές τοποθετήσεις, τις ακούσατε άλλωστε και φαντάζομαι είχα την αίσθηση ότι υπάρχει πολλή υποστήριξη προς το κλάδο του τουρισμού και εδώ είμαστε όλοι ενωμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα βλέπω ότι ε, η πρόσφαση Επιτροπή σημειώνει τα όσα υπόθηκαν ε, και σε σχέση με τον ε, προϋπολογισμό και σε σχέση με τις ε, δραστηριότητες. Κυρία Επίτροπε, μέχρι στιγμής μας δώσετε την υποστήριξή σας. Ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να το κάνετε και στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα ακούσατε πολλές παρεμβάσεις, πολλές ερωτήσεις και περιμένουμε με ανυπομονησία την απάντησή σας. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, πράγματι τέθηκαν πολλές ερωτήσεις ε, βεβαίως ξεκαθάρισα ήδη στην αρχή ότι θα σας δώσω σε όλους απαντήσεις γραπτά. Καταρχήν αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι εγώ δεν είμαι απεσιόδοξη για το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Αυτή είναι σταθερή μου πεποίθηση. Δεύτερον, είμαι επίσης πεπισμένη ότι αυτό, ότι ήρθε ο χρόνος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που έχουμε ένα πραγματικά περισμένο φάσμα νομικών εργαλείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί όπως απόθηκε εδώ, ε, πρόκειται κυρίως για μια εθνική τοπική περιφερειακή αρμοδιότητα. Ωστόσο, όλες σας οι παρατηρήσεις και οι παρεμβάσεις σας δείχνουν ότι πρωτίστως από τη δική μου οπτική γωνία δεν υπάρχει καμία ε, απόκληση. Και θα ξεκινήσω να εργάζομαι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή είναι η, το, αυτό είναι, αυτή είναι η αποστολή μου. Όπως το είπατε, πράγματι δεν αναφέρεται ο τουρισμός στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ανύπαρκτος. Βεβαίως υπάρχει και έχουμε πολλές ε, και παρόλο που εκφράζονται ε, κάποιες ανησυχίες για το ότι γίνεται ρητή μνήμα στον τουρισμό. Εγώ μπορώ να εξαγγείλω από τη δική μου σκοπιά και θα προσπαθήσω να πείσω και τα άλλα μέλη της Επιτροπής ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια νέα πρωτοβουλία. Ε, δεν, θέλω, δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί, έχουμε μια στρατηγική ε, και στο τέλος της εντολής μου θα ήθελα να υπάρξουν απτά αποτελέσματα, ίσως ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές. Όχι νέοι κανονισμοί, δεν είμαι θαυμάστρια των πολλών, οπαδός των πολλών κανονισμών, αν ίσως κάποιες νέες κατευθυντήριες γραμμές ή κάποια ανταλλαγή κοινών, ε, ε βέλτιστων πρακτικών, ή έστω ένα εγχειρίδιο εν σχέση με τη χρηματοδότηση, γιατί εδώ τέθηκαν και πολλές ερωτήσεις, αλλά το είπα αυτής εξ αρχής ότι το σχέδιο Juncker αφορά και τον τουρισμό. Ένα τέταρτο των, των χρημάτων πάει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρακτικά πολλά λεφτά. Και βεβαίως ο τουρισμός δεν έχει μια ξεκάθαρη διακριτή γραμμή, δεν ξεχωρίζει εμφανώς από, τον, από τις επιχειρήσεις. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει μια διευκρίνηση γιατί δεν είναι πολύ ξεκάθαρο για τις ε, τουριστικές επιχειρήσεις ε, πώς να αποτα... πού να αποτανθούν για να πάρουν τα χρήματα, πώς να υποβάλουν τις αιτήσεις κλπ. Όπως σας είπα υπάρχουν κάποιες ε, πηγές χρηματοδότησης, υπάρχουν τα διαστατικά ταμεία και εγώ ίδια προσωπικά είδα πολλές περιπτώσεις ε, χρηματοδότησης τουριστικών προγραμμάτων. Έχουμε το Ταμείο Κόσμε, ε, το οποίο, το οποίο διευθύνει η Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη. Ε, αλλά πολύ ξεκάθαρα αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι σωστή ενημέρωση. Με το εγχειρίδιο πού, μπορεί, πού θα πρέπει να αποταθεί κανείς για να βρει χρηματοδότηση για, το, για την επιχείρησή του. Βεβαίω ε, θα υπάρξει μια ευρεία διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα υπάρξει μια... Έχω κατά νου, όπως είπα, αυτή τη νέα πρωτοβουλία, ένα νέο πρόγραμμα δράση. Υπάρχει μια πολύ καλή βάση γι' αυτό και σίγουρα θα αποτελέσει μια σημαντική πηγή έμπνευση. Το τουριστικό μανιφέστο από την... Ε, υπό το πρίσμα του κλάδου. Και Πιστεύω ότι είναι η ενδεδειγμένη χρονική στιγμή. Α, και μπορούμε να δώσουμε 18 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών, αλλά ήδη τις προσεχείς εβδομάδες θα έχουμε τα πρώτα κείμενα, την πρώτη βάση ε, διαλόγου. Ε, βεβαίως το θέμα των δεξιοτήτων είναι πολύ καθοριστικό. Συμμετείχα τελευταία σε πολλές ε, σε διασκέψεις, σε διάφορους ε, κλάδους. Και το ζήτημα βέβαια της ψηφιοποίησης του, κλάδου, το θέμα των δεξιοτήτων ε, είναι πολύ καθοριστικά θέματα καθώς και η συνεργασία μεταξύ των πανεπιστήμιων, ή εκπαιδευτικών οργανισμών θα είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη σε αυτό το τομέα. Συνεργαζόμαστε στενά ε, με την Γενική για τις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να οικοδομήσουμε στη βάση αυτό που υπάρχει. Το ίδιο με την προσβασιμότητα στον τουρισμό και με τους αναπήρους υπάρχει μια καλή βάση για την μελλοντική μας εργασία. Το ίδιο ισχύει και για τον τουρισμό υγείας και τουρισμό των ΣΠΑ που είναι πηγή πλούτου για πολλές ευρωπαϊκές περιοχές και θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Όσον αφορά δε, το Ευρωπαϊκό Σήμα Ποιότητας, Υπήρξε μια πρόταση από την πλευρά της Επιτροπής πριν από μερικά χρόνια, αλλά δεν συμφώνησε το Συμβούλιο. Εμείς εδώ δεν έχουμε κάνει κάποια νέα πρωτοβουλία, ίσως όμως θα πρέπει να το κάνουμε, να το προσπαθήσουμε και πάλι. Αλλά ενδεχομένως είναι και δική σας ε, αρμοδιότητα, δικό σας ρόλος να πείσετε τις χώρες μέλη και το Συμβούλιο να δεχθεί την ιδέα αυτή του Ευρωπαϊκού Σήματος Ποιότητας στον τουρισμό. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία ανέφερα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τμήμα της συνεργασίας μας τους προσεχείς ε, μήνες καθώς και το sharing economy. Θα γνωρίζετε ότι αυτό είναι ένα από τα μείζωνα θέματα ε, στο οποίο έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα στην ενία ευρωπαϊκή αγορά. Ένα από αυτά είναι η συνεργατική οικονομία, το όπου τα αποτελέσματα είναι ορατά στον κλάδο των νοσοκομείων. Ε, είμαι πεπισμένη και ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει ένας νέος κανονισμός, αλλά θα πρέπει να ενοποιήσουμε τις προσεγγίσεις σε όλες τις χώρες μέλη. Δεν... Ε, και είδα μια πολύ καλή έκθεση από τις τουριστικές οργανώσεις. Νομίζω πέρσι ήταν το καλοκαίρι στη συνάντησή τους και πραγματικά άκουσα μια πολύ καλή παρουσίαση εδώ. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, θα πρέπει να ψάξουμε νέες ευκαιρίες σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα γιατί δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτό, είτε το θέλετε είτε όχι. Θα υπάρξουν αυτά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και θα αυξάνονται συνεχώς στο μέλλον. Ε, όπως σας είπα στην αρχή, ε, αποτελεί μια από τις δεσμεύσεις της ε, στρατηγικής ενίας αγοράς. Τα, ε, γύρω στα τέλη Ιουνίου θα παρουσιάσουμε λεπτομεριακές κατευθυντήριες γραμμές πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η φυστάμενη νομοθεσία γιατί θα πρέπει να είμαστε απολύτως εξασφαλμένοι για τα εξή τρία. Πρώτον, οι εταιρείε αυτές θα πρέπει να πληρώνουν φόρους. Δεύτερον, θέματα ασφαλείας των καταναλωτών. Τρίτον, ε, το θέμα του σήματος. Ε, εάν έχουμε καλές κατευθυντήριες ε, γραμμές και από την υφιστάμενη νομοθεσία, νομίζω ότι μπορούν τα πράγματα να λειτουργήσουν. Δεν είναι δυνατόν ε, τα μισά, οι μισές χώρες να καλωσορίζουν αυτές τις συνεργατικές μορφές οικονομίας και άλλες να τις απαγορεύουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και όπως σας είπα, αυτή είναι μια δέσμευση της, ενίας, για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και θα παράσχουμε στις χώρες μέλη όλα αυτά τα στοιχεία την άνοιξη, τέλος της άνοιξης. Τώρα, για την ε, επίδραση της ε, προσφυγικής κρίσης που ναι, είναι αρκετά νοπά τα πράγματα ακόμη και οι υπηρεσίες μας παρακολουθούν πολύ στενά το θέμα. Ε, παρακολουθούμε τα άμεσα, τις άμεσες συνέπειες προς το παρόν. Μπορούμε να σας δώσουμε, δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά μπορούμε να σας ε, δώσουμε και κάποια αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων που έχουμε κάνει για το πώς επηρεάζεται δηλαδή ο τουρισμός από την προσφυγική κρίση. Αλλά ε, να κλείσω λέγοντας ότι αυτά είναι τα ε, θέματα που... Α, ναι, ναι, έχουμε και, τα, έχουμε και τα ποδήλατα. Τα ποδήλατα, συγγνώμη, τα ποδήλατα. Ναι. Όχι, όχι, δεν είναι ρωτώ αλλά ξέρω και από τη δική μου την εμπειρία ότι πρέπει να υπάρχει στήριξη από τις περιφέρειες, γιατί υπάρχουν κονδύλια για να δοθούν σε ποδηλατόδρομους και στην Ανατολική Πολωνία είδαμε πολύ ωραία παραδείγματα κατασκευής ε, χιλιόμετρα, χιλιόμετρων ε, συγγνώμη, πολυδηλατόδρομων. Υπάρχουν τα κονδύλια, αλλά πρέπει να υπάρχει στήριξη από την, από την περιφερειακή κοινότητα. Δεν πρόκειται να πάει η Κομισιόν να χτίσει, να κατασκευάσει ποδηλατόδρομους. αυτό μπορεί να είναι ένα κομμάτι λοιπόν της ανάλυσης μας και του σχεδίου δράσης μας. Αλλά να σας πω το εξή. Είπα ότι θα σας ε, στείλουμε ένα concept paper, το οποίο θα είναι σύντομο, Και βεβαίως θα έρθουμε σε διαβούλευση, σε επαφή με τους εταίρους μας τον κλάδο, με τα μέλη του Κοινοβουλίου, με τις περιφέρειες, με τις κυβερνήσεις. Αλλά αν θα μπορούσατε κι εσείς ίσως να σκεφτείτε αυτό το μελλοντικό έγγραφο με τον τρόπο με τον οποίο το σκέφτομαι εγώ. Να είναι δηλαδή κάτι που δεν θα είναι πολύ εκτεταμένο, πολύ ευρύ, αλλά που θα έχει πραγματικά απτούς στόχους. Να έχουμε δηλαδή κάτι μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια που να μπορεί να πραγματοποιηθεί. Γιατί ήδη χρειάζεται μισή χρόνο, α πούμε, για να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Για να καταφέρουμε τελικά να κάνουμε πράξη τις ιδέες που θα περιλαμβάνει αυτό το concept paper. Νομίζω ότι ένα από τα θέματα που με απασχόλησαν εμένα είναι αυτή η σύνδεση με τη, μεταξύ της, των δημιουργικής, της δημιουργικής βιομηχανίας, το, της μόδας, του τουρισμού. Μπορούμε να, να προκύψουν και άλλες. Και έτσι θέλω να έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο κείμενο που θα μπορούμε να το μοιραστούμε και με τα κράτη-μέλη στο τέλος. Βεβαίως η πτυχή η οικονομική είναι πάρα πολύ σημαντική και οι πληροφορίες είναι φτωχές ε, βλέπω ότι πολλοί το λέτε ότι δεν υπάρχουν σωστές αξιόπιστες πληροφορίες ε, και οι τουρίστες δεν μπορούν ε, να βρουν που ακριβώς υπάρχουν σύνδεσμοι για δυνατότητες χρηματοδότησης. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα εγχειρίδιο σχετικά. Γιατί τα κονδύλια υπάρχουν, υπάρχουν πολλά λεφτά. Αλλά δεν είναι προφανές το πού βρίσκονται και δεν είναι καταγεγραμμένα ότι αυτά τα κονδύλια, τα τάδε θα πάνε στον τουρισμό. Οποιοδήποτε μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Οπότε πρέπει να ενημερώσουμε καλύτερα τους πολίτες για το πού μπορούν να βρουν τέτοιες δυνατότητες χρηματοδότησης. Ε, χάρηκα για την σημερινή συζήτηση που είχαμε. Εγώ θα σας στείλω τις ε, λεπτομέρειες και τις απαντήσεις ακόμη πιο λεπτομερώς και γραπτός και δεν θέλω να υπάρχουν κενά έτσι μεταξύ μας, θέλω να κάνουμε κάτι από τη θέση που είμαστε με τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Αλλά θέλω κάποιο, ένα αυτό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας, ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Βεβαίως ο τουρισμός και η ε, μετακίνηση ε, είναι, κοινές, είναι κοινά αντικείμενα στη δική μας την ε, Επιτροπή. Ελπίζω να μην, κρατήσει, να μην κάνουμε τρία χρόνια να σας ξαναδούμε στην Επιτροπή μας. Ελπίζω σύντομα να σας ξαναδούμε εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ.